Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Επειδή ο Πρόεδρο τη Επιτροπή είναι άρρωστο, ε, και ε, οι αντιπρόεδροι δεν μπορούν να παρευρεθούν, έχω και άλλη μια φορά σήμερα την τύχη να υποδεχτώ τους συναδέλφους και συναδέλφες καθώς επίσης και τους προσκεκλημένους μας και το θέμα αφορά την, ε, τις ενεργές πολιτικές ε, για την αγορά εργασίας των κρατών μελών, καλές πρακτικές όσον αφορά τα τρία μέρη της ε, στρατηγικής ε, για την ενεργό ένταξη, δηλαδή επαρκές εισόδημα, ενεργοποίηση της αγοράς εργασίας και υψηλές ποιότητες, ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες. Χαίρομαι ιδιαίτερος που έχουμε ειδικού καλεσμένους μεταξύ μα Ο καθένας από αυτού τους καλεσμένους θα μιλήσει 10 με 12 λεπτά, θα δώσει ε, τα σχόλιά του και θα παρουσιάσουν ε, και ε, τις παρουσιάσεις τους PowerPoint, τις οποίες μπορείτε να δείτε. Καλωσορίζω όλους τους καλεσμένους ε, την κυρία Λόλα Σαντιγιάννα Βαλέχο γραμματέα πολιτικών απασχόλησης ε, και μετανάστευσης ε, από την Ισπανία, την Καταλίνα Αλμάχο. Επίσης καλωσορίζω τον καθηγητή Γιάτσεκ Μέτσινα από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ε, του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας ο οποίος είναι ε, διευθυνών σύμβουλος ε, στην στον Πολωνικό Σύνδεσμο Λεβιάταν. Καλωσορίζω τον Πολ Σουέμ, ο οποίος είναι ανώτερος αναλυτής αγοράς εργασίας από τον ΟΑΣΑ και τον Λουκ Σέλντενο, ε, Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρόχων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία και τελευταίος αλλά όχι έσχατος, ο κύριος Στίβεν Τόμπιν, Διευθυντής Ομάδας ε, της ε, Μονάδας Αξιολόγησης Πολιτικών στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Καλώς ήρθατε. Και θα ξεκινήσουμε με την κυρία. Έχετε το λόγο. Ε, Καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση στην Επιτροπή Απασχόλησης Είμαι από την Καστήλια Λαμάντσα και από το Συνδικάτο το Ισπανικό. Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ώστε να συμπεριληφθούν τα άτομα που κανονικά αποκλείονται από την αγορά εργασίας λέει ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ελάχιστο εγγυημένο ποσό εισοδήματος στις ε, αγορές εργασίας και μαζί με ορισμένε υπηρεσίες πραγματικά ποιοτικές. Διακόπτη η ομιλήτρια. Στην Ισπανία έχουμε το ε, ελάχιστο εισόδημα από τις διάφορες αυτόνομες περιφέρειες, ε, το ελάχιστο ποσό εισόδημα μπορεί να έχει κανείς ε, και είχαμε ένα πρόγραμμα για την απασχόληση ώστε να συμπεριληφθούν εκείνοι που αποκλείται από την αγορά εργασίας και επίσης με την Δημόσια Υπηρεσία απασχόλησης και είναι αυτό μια αρεστή εικόνα πώς θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τη σύσταση της Επιτροπής την Ευρωπαϊκή σύσταση. Αλλά η πραγματικότητα ποια είναι. Πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμο στην Ισπανία είναι άνεργα πάνω από 2 χρόνια, από μακρύ χρονικό διάστημα δηλαδή. Και το 2011 είχε αυξηθεί ο αριθμό αυτός ε, κατά ένα εκατομμύριο ήδη. Αν κάνουμε μία ανάλυση σε κάθε αυτόνομη περιφέρεια τα εισοδήματα αυτά παρατηρούμε πώς η αγορά εργασία μας και η κοινωνία μας ε, έχει έρθει σε καινούργια επίπεδα φτώχεια. Υπάρχει ο καινούριο όρο ο φτωχό εργαζόμενο. Υπάρχουν ε, διαφορές ανάμεσα σε κάθε περιφέρεια και περισσότερα άτομα παίρνουν αυτά τα χρήματα αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ίσως ο αριθμός με όσους εκείνους αποκλείονται κοινωνικά και που έχουν ανάγκη. Πρόκειται για μια, ένα χαρακτηριστικό ότι αυτό συμβαίνει και σε περιφέρειες που έχουν ε, λιγότερους άνεργους. Αυτές οι περιφέρειες δίνουν περισσότερα χρήματα ενώ εκείνες που είναι φτωχότερες και κανονικά θα έπρεπε να βοηθάνε δίνουν λιγότερα, προσφέρουν λιγότερα χρήματα. Και ακόμα κάτι Έχουμε και το άλλο σκέλος. Ποιο είναι αυτό. Είναι οι πολιτικές απασχόλησης και οι περικοπές οι οποίες συμβαίνουν σε αυτές τις πολιτικές απασχόλησης. Τα δύο κάθε από κάθε τρία ευρώ θα έπρεπε κανονικά να τα επενδύει για την ε, αγορά εργασίας. Έχουμε ένα ελάχιστο ακριβώς εισόδημα για να μπορέσουν να συμπληρωθούν τα άτομα στην αγορά εργασίας. Κάτι ακόμα που παρατηρούμε είναι ότι η κυβέρνηση ήρθε σε αντίθετη κατεύθυνση με εκείνη που πρότειναν η Επιτροπή και η Ευρώπη γενικά. Βλέπουμε ότι είχαμε να αφορούνται εκεί που υπάρχουν λιγότερες επιχειρήσεις, εκεί δίνονται λιγότερα χρήματα, εκεί έγιναν οι περισσότερες περικοπές. Και όπως το βλέπουμε εδώ στο γράφημα, στο Καστίλια Λαμάντσα, είχαμε 90% μπορούμε να πούμε περικοπές από από τα 85 κάπου ευρώ που δινόταν, προσφερόταν. Έχουμε μόνο 40 από εκεί και πέρα. Και έτσι βλέπουμε ότι εκεί που έχουν τις περισσότερες επιχειρήσεις, εκεί είχαμε τις λιγότερες περικοπές. Παράδεξο. Ε, το αντίθετο από αυτό που υποδεικνύουν οι κατευθυντήριες γραμμές και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι σημαίνει αυτό, ότι ήταν μια διαβολική μηχανή αυτή η στρατηγική και έχουμε συνδικάτα που συμφώνησαν στις απολύσεις ε, πιο εύκολες ε, και πολλά πράγματα, πολλές παροχές μειώθηκαν ταυτόχρονα όμως και δραστήριες πολιτικές απασχόλησης και η κυβέρνηση μαζί με τα συνδικάτα βλέπουμε ότι ασχολούνται με αυτό, αλλά δυστυχώς τα πράγματα χειροτερεύουν και δεν σέβονται τις ευρωπαϊκές συστάσεις. Ένα ελάχιστο εισόδημα μαζί με μια παρακολούθηση αυτών των πληθυσμών που έχουν φύγει και αυτό που συνέβη είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις που απαιτούνται σε πολλές περιπτώσεις και συνεχίζουν πάντα να ισχύουν για να μπορέσει κανείς να υποφεληθεί από αυτό το εργαλείο και όταν πάνω από 330.000 άτομα πούμε που θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα 400 τόσα ευρώ ε, θα δυστυχώ δεν διαθέτουν τι προποθέσει. δεν πληρούν τι προποθέσει και οι 313.000 γίνονται 31.000 τελικά. Οι άλλοι αποκλείονται. Όπως έχει σήμερα το πρόβλημα είναι ότι αυτέ οι προποθέσει οι απαιτήσει είναι ιδιαίτερα υψηλές, πολλά εμπόδια και ουσιαστικά αποκλείονται. Και επιμένει κανείς για ορισμένα συνοδευτικά μέτρα, αλλά δεν υπάρχει η απαραίτητη βοήθεια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και η δημόσια υπηρεσία χειροτερεύουν οι προσφορές της, οι παροχές της ε, λόγω αδυναμίες. Βλέπουμε λοιπόν τους άνεργους να υποφέρουν, τους νέους να υποφέρουν που ξέρουμε ότι περίπου το 60% των νέων είναι άνεργο και στην αρχή έλεγαν για μία εγγύηση αυτούς τους νέους, αλλά πέτυχε παταγωδός γιατί εκεί που πήγαινε αυτή η βοήθεια δεν πήγε πραγματικά και δεν υπήρξαν τα κατάλληλα συστήματα για να επιτευχθεί αυτό. Εμείς έχουμε μία πρόταση για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Είναι ένα πρότυπο κοινωνικού διαλόγου μαζί με τα συνδικάτα, μαζί με την κυβέρνηση για να κάνουμε μία εκτίμηση για αυτές τις αποκλήσεις, για αυτές τις παρεκκλήσεις στην εφαρμογή αυτών των σχεδίων που ουσιαστικά είναι μόνο μια βιτρίνα προς τα έξω για να δείξουν ότι δήθεν κάνουν πράγματα αλλά κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει για όλα αυτά τα άτομα τα οποία είναι αποκλεισμένα κοινωνικά να μπορέσει να υπάρξει αυτό το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις, σε μια ενεργό πολιτική και να υπάρξει μια επένδυση με περισσότερους πόρους από το δημόσιο και ταυτόχρονα μια σαφής αύξηση των δραστηριοτήτων δικαστήριων πολιτικών απασχόλησης για να φτάσουμε και πάλι στο επίπεδο του 2008 σύμφωνα και με τις κατευθυντές γραμμές των Βρυξελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δαπάνη που θα πρέπει να γίνεται ώστε όλοι εκείνοι που είναι απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας που θα πρέπει να έχουν τα μέσα για να ανταπεξέλθουν, να μπορέσουν να εταχθούν σε αυτές τις αγορές να γίνει πραγματικότητα αυτή η ένταξη. Εμείς πραγματικά ανησυχούμε, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Θέλουμε να πάμε κάπως ε, πιο πέρα από τα εμπόδια που θέτουν οι κυβερνήσεις και από τα σχέδιά τους όπως αυτό το πρόγραμμα και να μπορέσουν αυτά να αποτελέσουν κάτι το αποτελεσματικό και το βλέπουμε, βλέπουμε τις συνθήκες που ισχύουν στις χώρες, στη χώρα μας ε, βλέπουμε ότι δυστυχώς υπάρχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που εύχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και για τη δική μας δουλειά και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον καθηγητά Γιάτσεκ Μέτσινα. Μπορείτε να με διορθώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επικεντρωθώ ε, στις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει η Πολωνία τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την αγορά εργασίας που δεν αποκλείει. Η βάση της ανάλυσης μου είναι, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι όταν η Πολωνία έγινε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή πριν 10 χρόνια, είχε την υψηλότερη ανεργία αλλά και τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης. Αγωνιστήκαμε με την ανεργία και το καταφέραμε, όμως ε, είχαμε και μια άλλη πρόκληση τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή θέλαμε να εκμεταλλευτούμε το εκμετάλλευτο ε, προσωπικό και πώς θα το κάνουμε αυτό. Εδώ έχουμε τέσσερις ομάδες, ε, τους άνεργους, ε, κατά 50% είναι μακροχρόνια άνεργοι αλλά και πάρα πολλοί νέοι καθώς επίσης και πολλές άνεργες γυναίκες. Η δεύτερη ομάδα τώρα είναι άτομα τα οποία εργάζονται μονάχα σε καθεστώς μερικής απασχόλησης καθώς επίσης και άτομα τα οποία δεν απασχολούνται όπως επίσης και αυτοί οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας αλλά και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τη βούληση να επιστρέψουν. Όλα αυτά δείχνει λοιπόν ότι το 16% μπορεί να αυξηθεί η δυνατότητα απασχόλησης στην Πολωνία αν επικεντρωθούμε στις δύο ομάδες. Πρώτον, οι άνεργοι, το βασικό πρόβλημα είναι οι νέοι Αυτά είναι στοιχεία από το 2012, αυτή ήταν η βάση μας όταν το 2013 και 2014 πραγματοποιήσαμε μεταρρυθμίσεις. Πρόκειται λοιπόν για νέους ανθρώπους, ε, γυναίκες, που, έχουν, ε, που δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, αλλά και αυτοί οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι ε, των 50. Γενικότερα η κατάσταση έχει ως εξής αυτοί ε, είναι λοιπόν καταρτισμένοι, δεν έχουν επαρκή κατάρτιση και για αυτόν τον λόγο υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της ανεργίας. Η δεύτερη ομάδα πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν κανένα κίνητρο να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και σε αυτό το τομέα λοιπόν θα θέλαμε να επικεντρωθούμε ιδιαίτερως στους μεγαλύτερους σε γυναίκες που ε, έγιναν μητέρες και στη συνέχεια δεν επιστρέφουν στην αγορά εργασίας. Η συγκεκριμένη ανάλυση λοιπόν ήταν για εμάς μία βάση πάνω στην οποία μεταρρυθμίσαμε την αγορά εργασία μας και εδώ έχουμε τέσσερις διαφορετικούς τομείς που μας ενδιαφέρουν ε, μία ε, διαχείριση των κρίσεων με τη δημιουργία ε, προφίλ για αυτούς τους ανέργους, στη συνέχεια διάφοροι δείκτες τους οποίους έχουμε δημιουργήσει καθώς επίσης και νέα μέσα. Έχουμε αρκετά νέα μέσα τα οποία τα δημιουργήσαμε για αυτό το σκοπό και ιδιαιτέρως για να δοθεί η πρόσβαση στους νέους στην αγορά εργασία, δηλαδή ανθρώπους κάτω της ηλικίας των 30, αλλά και για αυτούς που είναι άνω των 50, καθώς επίσης και οι γυναίκες είναι μια τρίτη ομάδα στόχος. Το θέμα λοιπόν είναι να τους προσφέρουμε εργασία και ταυτόχρονα να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας η ε, δομή της δημόσιας απασχόλησης στην Πολωνία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα, έχουμε, πολύπλοκη, έχουμε διάφορα επίπεδα. Και εδώ λοιπόν έχουμε δυνατότητες να δημιουργήσουμε αυτές τις εταιρικέ σχέσεις ε, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ενώ ταυτόχρονα έχουμε την ε, δυνατότητα να κινηθούμε καθαρά δημόσια ή δημόσια κοινωνικά το οποίο σημαίνει οι υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να απασχοληθούν έτσι ούτως ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές ε, ενώ ταυτόχρονα δημιουργήσαμε και ένα, ε, μια, ε, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο οι κοινωνικοί εταίροι το χειρίζονται από κοινού. Τόσο οι εργαδότες δηλαδή όσο και οι εργαζόμενοι. Επιπρόσθετα μέσα εμείς τα κάναμε πιο χαλαρά. Αυτό χρηματοδοτείται και από τους ε, εργοδότες όμως ε, έχουμε ε, πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και όλο αυτό έχει πάρα πολλά καλά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταφέρουμε να αποφύγουμε αυτό το κίνδυνο, αυτό το ρίσκο και να επικεντρωθούμε στις αγορές εργασίας οι οποίες ε, στην προκειμένη περίπτωση ασχολούνται κυρίως στο να δώσουν κίνητρα προς τους ανέργους. Όμως επιπρόσθετα αυτό που θέλουμε είναι να προσεγγίσουμε και αυτούς οι οποίοι απέχουν πάρα πολύ από την αγορά εργασίας ε, τόσο ε, το οποίο το επιτυγχάνουμε τόσο από, ε, ε, από την ίδια την αγορά εργασίας όσο και με ΜΚΟ και έτσι λοιπόν καταφέραμε ε, να επιτύχουμε κάποια αποτελέσματα και σε αυτό το τομέα. Αλλά και το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι ένα κεντρικό πρόγραμμα και στις επιχειρήσεις, στους εργοδότες. Εδώ οργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα. Αναλάβαμε το 100% των κόστων για τις μικροεπιχειρήσεις Κατά το πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το συγκεκριμένο ταμείο, πάνω από ε, χίλιοι εργοδότες το χρησιμοποίησαν, ενώ εμείς ως ε, Πολωνία έχουμε γενικότερα δυσάρεστα αποτελέσματα όταν το ζήτημα αφορά τη διαβίου μάθηση, οπότε πιστεύω ότι σε αυτό το τομέα μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα. Επιπλέον έχουμε και άλλους τομείς στους οποίους εργαστήκαμε όπως ε, συνεργασίες με τους εργοδότες ενώ συνδυάσαμε τη χρηματοδότηση με το δημόσιο τομέα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν ε, τις επιχειρήσεις ε, δεν θα πρέπει να πηγαίνουν προς την κατεύθυνση των αποφύτων αλλά των φοιτητών οι οποίοι σπουδάζουν ακόμα και πρακτικά βρίσκονται λίγο πριν την αποφύτησή τους. Όσον αφορά τώρα τη συνεργασία με τους εργοδότες, εκεί εισάγαμε νέες δομές management, δηλαδή κάθε νέος ο οποίος έχει το κίνητρο μπορεί να λάβει μια τέτοια δυνατότητα και κάθε τέτοιο άτομο μπορεί να λάβει τη δυνατότητα να κάνει μια πρακτική άσκηση από κάποιον εργοδότη και έτσι στη συνέχεια μπορούν να ε, προσληφθούν από τους ε, εργοδότες οι οποίοι οι ίδιοι τους έχουν αναζητήσει. Βέβαια δεν είναι πάντοτε επιτυχές, όμως ε, παρόλα αυτά έχουμε τους αντίστοιχους συμβούλους οι οποίοι ενημερώνουν και προστατεύουν τους νέους από το 2014 δηλαδή, από τότε που έγινε η συγκεκριμένη αλλαγή στην ε, αγορά εργασίας ή τα ποσοστά απασχόλησης εκτινάχθηκαν στα ύψη, το οποίο όπως είπα ε, και πριν ε, για την Πολωνία είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και βλέπουμε μια τάση όπως φαίνεται στο κάτω γράφημα ότι η απασχόληση αυτή, η τάση αυτή λοιπόν είναι αυξητική Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η Πολωνία ανήκει στις χώρες όπου τα ποσοστά ανεργίας μειώνονται, έχει μια πάρα πολύ καλή ε, δυναμική. 7,1% όμως κάτι ακόμα η δομή της ε, πολωνικής ανεργίας αλλάζει και στο πλαίσιο των εγγυήσεων για την νεολαία έχει μειωθεί η ανεργία από το 28% στο 22,7% και νομίζω ότι φέτος θα μπορέσουμε να πέσουμε κάτω από το 20%. Προσπαθούμε επίσης να επέμβουμε και στην αγορά εργασίας όταν το ζήτημα αφορά ανθρώπους οι οποίοι είναι άνω των 50 ετών και εδώ λοιπόν προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης ούτω ώστε να ενισχύσουμε την ελκυστικότητα των ε, μεγαλύτερων ε, ανθρώπων το σημαντικό είναι ότι το ποσοστό ανεργίας στους μακροχρόνια ανέργους αυξάνεται και εδώ πράγματι λοιπόν θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο. Επιπλέον θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Πολωνία δεν προσπαθεί μονάχα να βελτιώσει την κατάσταση στην αγορά εργασίας, όμως ε, ταυτόχρονα έχουμε και μια άλλη ε, πρόκληση η οποία αφορά την τον έντονο κατακαιρματισμό της αγοράς ε, εργασίας ε, τον τελευταίο χρόνο αλλά και φέτος. Ε, ξεκινήσαμε ένα, ένα ταμείο και ταυτόχρονα κάναμε και συμβάσεις και προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε περισσότερα, ε, περισσότερες συμβάσεις περιορισμένου χρόνου ενώ ταυτόχρονα αρχίσαμε να επενδύουμε περισσότερο και στην ε, ε, οικογενειακή πολιτική όπως αφορά την ευελιξία για την άδεια εγκυμοσύνης ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε για παιδιά μέχρι ηλικίας των τριών ετών να υπάρχουν θέσεις ε, σε βρεοκφοκομεία, ολοήμερα βρεοκφοκομεία. Ενώ τέλος θα ήθελα να ε, αναφέρω κάτι ακόμα το οποίο ανάφερε και η ε, προηγούμενη ομιλήτρια. Είχαμε αυτή τη διεθνή κρίση και υπήρχαν εντάσεις και στην Πολωνία και είδαμε λοιπόν στην Πολωνία ότι υπήρξε ένας διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και τον Σεπτέμβριο λοιπόν δημιουργήσαμε μια νέα δομή, στόχος της οποίας είναι να προωθήσει την ευελιξία αλλά και την ασφάλεια ε, στην ε, αγορά εργασίας. Είναι μια μορφή την οποία ξεκινήσαμε πρόσφατα Συνοπτικά λοιπόν έχουμε περισσότερους δείκτες αποδοτικότητας, μπορούμε πράγματι να δράσουμε πάνω στην αγορά εργασίας και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για διάφορες συνεργασίες δημόσιες και ιδιωτικές για παράδειγμα αλλά και τις άλλες ε, συνεργασίες. Χάρη λοιπόν σε αυτές τις ε, συνεργασίες διευκολύνεται το έργο μας στην αγορά εργασίας. Επιπλέον αυτές ε, οι δράσεις έχουν ως αποτέλεσμα η ποιότητα της εργασίας να αυξάνεται και περιορίζουν αυτόν τον κατακαιρματισμό στην αγορά εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα περάσουμε στον επόμενο ομιλητή. Πολ Σουέιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη μου χαρά εκ μέρους των συναδέλφων στον ΟΣΑ με τους οποίους δουλεύουμε για τις ε, κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησεις να σας παρουσιάσω το, δική μας, το δικό μας προβληματισμό για το πώς βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ενεργή εργοένταξη και πώς θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο επιτυχημένη από ό,τι σήμερα. Αυτό που θέλω να κάνω τα ερχόμενα λεπτά είναι να πω ποια ήταν τα δικά μου ατομικά διδάγματα από δύο φάσεις εργασίας που τελικά συνδυάσαμε στον ΟΣΑ, διότι νομίζω ότι από κοινού δείχνουν τι ρόλο μπορούν να παίξουν τα ενεργά προγράμματα για την αγορά εργασίας και πώς οι μη απασχολούμενοι και άνεργοι μπορούν να περάσουν σε θέσεις εργασίας πιο βιώσιμες. Πώς θα φέρουμε τους ανέργους στις θέσεις εργασίας λοιπόν είναι το ένα θέμα. Αυτοί που προσφάτως έχουν χάσει τη δουλειά τους πολλές φορές είναι στην ίδια θέση με αυτές που είναι πιο πολύ καιρό εκτός αγοράς εργασίας. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η δική μας προσέγγιση να αλλάξει πολύ. Εκεί που αλλάζουν επίση πολύ τα πράγματα στο να διακρίνουμε ομάδε ανέργων είναι οι αναπηρίε, κάποιο φυσικό ελάττωμα και εκεί αλλάζει το στοιχείο τη ένταξη στην αγορά εργασία. Πρώτα απ' όλα, να σας παρουσιάσω τη δική μας συλλογιστική, πώς ε, μπορούμε να έχουμε ενεργό πολιτική, ενεργοποίηση για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Μία μορφή πιο συμμετοχική που να οδηγεί στη συμμετοχή όλων. Τέσσερα στοιχεία χρειάζονται. Τα τρία είναι οι λειτουργικές ε, ανάγκες του συστήματος και το τέταρτο είναι το πώς ε, συνδυάζονται όλες αυτές οι ανάγκες μεταξύ τους. Πρώτη ανάγκη είναι να βεβαιωθούμε ότι όσοι δεν εργάζονται έχουν κίνητρα και ενθαρρύνονται να ε, δουλέψουν για να ψάξουν δουλειά. Ήδη αναζήτηση εργασίας για κάποιους είναι ένα θέμα, αλλά υπάρχουν πολλοί που χρειάζονται στήριξη για να ξεπεράσουν φραγμούς ώστε να φτάσουν επιτυχώς στην αγορά εργασίας. Μια από τι προποθέσει για να πετύχει κανεί είναι να υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα. Να πιστεύουν ότι μπορεί να πετύχουν κάτι και έτσι να επωφεληθούν από κάθε βοήθεια που μπορεί να τους προσφέρεται. Δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που ονομάζουμε απασχολησιμότητα. Για να τα πάει κανεί καλά στην αγορά εργασία πρέπει τους ε, ενδεχόμενους εργοδότες να παρουσιάζει υψηλή παραγωγικότητα σε σχέση με άλλους ε, απασχολούμενους. Αυτό δεν είναι έτοιμο να το προσφέρουν όλοι αυτοί αμέσως. Είναι θέμα δεξιοτήτων, ε, περαιτέρω εκπαίδευση, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλοι φραγμοί κοινωνικού τύπου, όπως το να είναι κανείς επιτυχής στη δουλειά του και παραγωγικός. Μετά είναι το θέμα του τι ευκαιρίες διαθέτουμε στους ανέργους ώστε να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά του, εφόσον έχουν κίνητρα να εργαστούν και να έχουν και εργοδότες λόγο να του προσλάβουν. Αυτά τα τρία στοιχεία πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ του και έτσι. Τα ενεργά προγράμματα για την αγορά εργασία δίνουν έμφαση κυρίω στο δεύτερο στοιχείο, την αυξημένη απασχολησιμότητα. Όμω, δεν θα υποφεληθεί κανεί πλήρω από τα ενεργά αυτά προγράμματα εάν δεν συνδυάσει και τα άλλα δύο στοιχεία. Για να συνδυαστούν λοιπόν χρειάζεται το θεσμικό πλαίσιο ώστε όλες αυτές οι λειτουργικές ανάγκες να καλύπτονται με έναν τρόπο συντεταγμένο. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να εξηγήσω το κάθε σημείο από αυτά ξεχωριστά και να προσπαθήσω να εξηγήσω τη συλλογιστική αυτών που έχουν ιδιαίτερου φραγμού ω προ την εργασία. Τι δυσκολίε αντιμετωπίζουν σε σχέση με κάποιον που λόγω χάρη έχει μια σταθερή θέση εργασία και, κάποια, και μια μεγάλη πείρα χάνει ξαφνικά τη δουλειά του, αλλά πολύ πιο εύκολα μπορεί να επανενταχθεί στην αγορά εργασία. Μα ενδιαφέρουν οι δυσκολότερε περιπτώσει. Ω προ τα κίνητα και την κινητοποίηση, λοιπόν, αυτό που συνήθω ε, τονίζει ο Σάκη είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν οικονομικά κίνητρα, δηλαδή να είναι ελκυστικό για κάποιον να επιστρέψει στην αγορά εργασία, δηλαδή το εισόδημα, ο μισθό, τα ωφελήματα που λαμβάνει. ο λόγο που θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να επιστρέψει στην αγορά εργασία θα πρέπει να είναι και οικονομικό. Όμω αυτοί που απέχουν περισσότερο από την αγορά εργασία ε, χωρίζονται σε δύο περιπτώσει. Ε, αυτοί μπορεί να έχουν αποθαρρυνθεί ιδιαίτερω από την αγορά εργασία γιατί δεν πιστεύουν ότι εκεί μπορούν να αντίσουν. Θα πρέπει λοιπόν να του δώσουμε και κάποια συμβουλευτική στήριξη. Και γιατί και για αυτούς υπάρχει στρατηγική που μπορεί να πετύχει για την ένταξή του στην αγορά εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστεί μαζί του κάποιο σύμβουλο, να ε, σχεδιάσει ε, ένα πρόγραμμα σε πολλά στάδια και το τελικό στάδιο να φτάσουν να αναζητούν εργασία, αλλά προηγουμένω να έχουν εντοπίσει ποια είναι τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν για, την... για να φτάσουν στην αγορά εργασία και αυτά να αντιμετωπιστούν πρώτα. Ερεσιμότητα τώρα και επιδόματα. Εκεί αφού υπάρξει συμβουλευτική δουλειά θα πρέπει να αξιοποιήσουν ε, τεχνικώς στα, τη στήριξη που τους έχει δοθεί για να ψάξουν για δουλειά. Έτσι θα σταθούν ελεύθεροι να ε, ψάξουν καλύτερα. Ως προς την απασχολησιμότητα. Αυτό κάνουν συνήθως τα μερικά προγράμματα για την αγορά εργασίας. Ε, εκπαίδευση, δεξιότητες, κάποιοι που έχουν μέση εκπαίδευση ή μετανάστες γλωσσική εκπαίδευση κάποιες φορές, τέτοιου είδους στόχοι προγραμματίζονται. Όμως αυτό που θέλω εγώ να τονίσω εδώ είναι ότι είναι σημαντικό αυτές οι μορφές στήριξης και βοήθειας να προσφέρονται στο πλαίσιο ενός γενικότερου προγράμματος. Δηλαδή να καταλαβαίνει ο ε, ενδιαφερόμενος αργότερα θα οδηγηθεί ε, στην αγορά εργασίας και μετά να βρει και μια κατάλληλη θέση όντως για να δει στην πράξη πόσο σε βελτίωσε τι δεξιότητέ του και δεν του πρόσφερε αυτό. Του πρόσφερε αυτό. Τρίτο σημείο τώρα, οι ευκαιρίε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε τι κατάλληλε ευκαιρίε για του ανθρώπου εφόσον βελτιώσουν ε, το ποσοστό απασχολησιμότητά του, εντοπίσουν τι μπορούν να προσφέρουν σε έναν μελλοντικό εργοδότη και μπορούν να αρχίσουν να αναζητούν δουλειά. Εδώ οι δημοσκοπήσεις για την ε, κρατική επασχόληση από το φορέα που συνήθως μας δίνει τέτοιου είδους στοιχεία και μεσολαβίως ως διάμεσος μεταξύ όσων αναζητούν εργασία και των ε, εργοδοτών, των επίσημων εργοδοτών, βλέπουμε ότι όσοι για ένα σχετικό διάστημα δεν έχουν εργαστεί μπορεί να έχουν και κάποιο άλλο θέμα ένα σωματικό ελάττωμα λόγου χάρη. Όμω αυτοί οι φορεί ακριβώ καταλαβαίνουν καλύτερα τις ανάγκες των εργοδοτών και μπορούν να φροντίσουν να κάνουν τους κατάλληλους διακανονισμού ώστε τα άτομα αυτά να βρουν τελικά δουλειά. Δηλαδή πρέπει να γίνει πρώτα μια συζήτηση μεταξύ του κρατικού φορέα για την απασχόληση και του ανθρώπου που αναζητά δουλειά για να επιληθεί το κάθε πρόβλημα σε ατομικό επίπεδο. Επίσης, μπορεί να υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο όπως παρακολουθούμενη εργασία που να λειτουργήσει ως ε, μέσο διάστημα μέχρι να βρουν μια μόνιμη θέση αυτοί που αναζητούν εργασία. Κάτι άλλο που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον στη δεύτερη διαφάνεια είναι να δούμε τι εμπειρία έχουμε σήμερα την υλοποίηση των ε, στρατηγικών ενεργούς ένταξης, ενεργού ένταξης. Εδώ, εκεί που υπάρχει μια διαφορά, είναι ότι συνήθως τα προγράμματα απασχόλησης υποτίθεται ότι είναι πολύ επιλεκτικά, δηλαδή ε, επιλέγουν αυτούς που είναι σχεδόν έτοιμοι να ξαναπεράσουν στην αγορά εργασίας όχι αυτούς που έχουν πραγματικά εμπόδια και δυσκολίες. Ως προς τους πόρους μας όμως, είναι σημαντικό να μην κάνουμε αντιπαράθεση μεταξύ των διαφορετικών ομάδων. Εάν πετυχαίνουμε καλά αποτελέσματα με αυτούς που έχουν υψηλά ποσοστά απασχολησιμότητας ε, και βρίσκουμε θέσεις, δουλειά, δουλειά, θέσεις για αυτούς πολύ γρήγορα, θα είναι αντιστρόφως ε, δυσκολότερο να βοηθήσουμε κάποιον που έχει μείνει εκτός ε, αγοράς εργασίας για πολύ καιρό. Είναι πολύ πιο εύκολο κάποιο που έχασε τη δουλειά του από ένα-δύο μήνε και έχει μεγάλη πείρα να ξαναβρει δουλειά από ότι κάποιο που έχει μείνει εκτό για μεγάλο διάστημα. Αυτοί λοιπόν είναι που μα ανησυχούν περισσότερο και αυτοί είναι που δυσκολότερα ε, προσλαμβάνονται ξανά από του μελλοντικού εργοδότε. Εδώ Πρέπει λοιπόν να δίνουμε βοήθεια όχι μόνο στις πιο εύκολες ομάδες, αλλά να φροντίζουμε να δίνουμε έμφαση και στους ε, μακροπρόθεσμα άνεργους. Και το αντίστροφο, επίσης εφόσον κάνουμε περισσότερα για τους προσφάτως άνεργους, μπορούμε να κάνουμε λιγότερα για όσους είναι περισσότερο καιρό άνεργοι. Τώρα για το τι θεσμική δουλειά μπορεί να γίνει εδώ. Τι μπορούν να κάνουν οι υπεύθυνοι φορεί. Οι υπηρεσίε ενεργού απασχόλησης Πολλέ φορές ασχολούνται με ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένα προβλήματα, γονεί που δεν έχουν εργαστεί πολλά χρόνια γιατί φρόντιζαν τις οικογένειέ τους, ανθρώπους με αναπηρίε και το καθεξή. Εδώ Κοιτάζοντας διαφορετικές χώρες, καταλήγω ότι το πρόβλημα δεν είναι ποιος αναλαμβάνει, εάν είναι ένας ο φορέας ή πολλοί αυτοί που φροντίζουν ε, την επαναπρόθεση των ανθρώπων ε, προς την αγορά εργασίας. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχουν και οι απαραίτητες ε, ειδικέ γνώσεις, εφόσον υπάρχουν ας πούμε, προβλήματα υγείας στους ανέργους. Κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Εκεί χρειάζεται να πάρουν μέρος και οι συγκεκριμένοι ειδικοί που θα δουν ε, με ιδιαίτερο τρόπο αυτά τα προβλήματα. Ο συνδυασμός λοιπόν είναι που ε, μετράει, γιατί έτσι το άτομο που χρειάζεται θα λάβει τη βοήθεια που θα τον βοηθήσει. Αυτά ήταν τα στοιχεία που ήθελα να αναπτύξω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, mm, Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πάουλ Σουέιμ. Θεωρώ ότι η ευθύνη και η δραστηριότητα ε, και το πώς μπορούν αυτά να βοηθήσουν ε, να μειώσουν ε, την ανεργία στην Ευρώπη. Θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να έρθω πιο νωρίς γιατί είχα άλλες υποχρεώσεις. Τον λόγο έχει ο κύριος Λουκ Λου. Ε, Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Παροχής Υπηρεσιών για Ανθρώπους με Αναπηρίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ε, που με προσκάλεσε για να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις και ιδέες σχετικά με πολιτικές για την εργασία καθώς επίσης και πολιτικές και δραστηριότητας ε, από όλη την Ευρώπη. Είμαι ο Γενικός Διευθυντής ε, της, ε, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου της Παροχής Υπηρεσιών για Ανθρώπους με Αναπηρίες. Εκπροσωπούμε πάνω από 11.000 οργανώσεις μέχρι στιγμής που είναι ενεργές σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περίπου το 1 τρίτο αυτών των οργανώσεων παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης όπως ε, για παράδειγμα ε, επαγγελματική κατάρτιση. Το θέμα αυτό λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς και όταν ε, κανείς με ρωτάει ποιος είναι ο συνολικός μας στόχος πάντοτε απαντάω λέγοντας ότι παρέχουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και με συνοχή. Στην σύντομη εμβέμβασή μου θα, ε, θα επικεντρωθώ σε δύο σημεία. Αρχικά θα κάνω γενικά σχόλια και στη συνέχεια θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ε, μερικά ευρήματα σχετικά με μια ανάλυση επιτυχίας που πραγματοποιήσαμε ε, σε σχέση με προγράμματα απασχόλησης. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσω με κάποια γενικά σχόλια και ανησυχίες Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να απομακρυνθούμε από το να κατηγορούμε τη γλώσσα τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε ακόμα. Έχουμε την τάση να μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ μακριά από την αγορά εργασίας, από, ε, οι οποίοι είναι απομακρυσμένοι. Και χωρίς λοιπόν να έχουμε αυτή τη βούληση, αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι ότι κατηγορούμε ανθρώπους επειδή δεν απασχολούνται, επειδή δεν εργάζονται και αυτό βέβαια τροφοδοτεί την ιδέα ότι η αγορά εργασίας είναι κάτι μονολυθικό, κάτι το οποίο δεν μπορείς να κατευθύνεις, κάτι που δεν μπορείς να διαχειριστείς. Αυτό λοιπόν το οποίο παρατηρώ με βάση τα επιτυχημένα προγράμματα σε όλη την Ευρώπη είναι ότι τα πιο επιτυχημένα είναι αυτά τα οποία δεν έργασε μονάχα με τους πολίτες αλλά και με, τους, ε, με τις επιχειρήσεις, με την αγορά εργασίας και προσπαθείς ε, να τροποποιήσεις ε, τα επαγγελματικά προφίλ, τις απαιτήσεις, για θέσεις εργασίας και έτσι λοιπόν προσπαθείς να συνδυάσεις όλα αυτά. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να απομακρυνθούμε από την γλώσσα αυτή. Η αγορά εργασία ή ε, εργοδότες χρειάζονται λοιπόν πάρα πολύ υποστήριξη για να μπορέσουν ε, να κάνουν πιο ε, περιεκτικέ τις επιχειρήσεις τους η συνέπεια της κρίσεως τώρα. Η κρίση όπως γνωρίζουμε δεν έχει τελειώσει και το ξέρουμε αυτό και από προηγούμενες κρίσεις. Ο κοινωνικός τομέας, ο ε, τομέας της υγείας, της εκμέδευσης είναι αυτός που προσβάλλεται περισσότερο και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με άλλους τομείς στην κοινωνία και σιγά σιγά αρχίζουμε να νιώθουμε τις συνέπειες των μέτρων λιτότητας το βλέπουμε αυτό ε, σε οικογένειες που έχουν κάποιο άτομο με αναπηρία, που έχουν χάσει ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδήματός τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμμετέχουν τόσο εύκολα στην κοινωνία, δεν έχουν πρόσβαση τόσο εύκολα στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα βλέπουμε και μια απώλεια στις υπηρεσίες ποιότητας. Οι περισσότερες λοιπόν υπηρεσίες που μπορούσαν να ξεπεράσουν τα μέτρα λιτότητας το έκαναν αυτό απολύοντας κόσμο. Οπότε λοιπόν υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι που είναι διαθέσιμοι ώστε να παράσχουν ε, υπηρεσίες υποστήριξης. Και πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα, ε, τα ε, πιο καινοτόμα μοντέλα ένα, για να μπορέσουν άτομα με αναπηρία να μπουν στην αγορά εργασίας τέτοιες υπηρεσίες και οργανισμοί έχουν υποστεί τα περισσότερα λόγω των μέτρων λιτότητας. Είναι λίγο περίεργο ότι ακόμα και μοντέλα τα οποία έχουν αποδείξει ότι φέρουν επιστροφές ένα προς 5 ε, για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται ε, ε, πέντε επιστρέφουν στην κοινωνία αυτά τα μοντέλα υποστήριξης είναι που υποφέρουν περισσότερο από την κρίση σε σχέση με άλλα. Οπότε Συνοψίζοντας το πρώτο μικρό μου κεφάλαιο, όσον αφορά την στρατηγική χωρίς αποκλεισμούς, όλα αυτά είναι σημαντικά. Η υποστήριξη εισοδήματος, δηλαδή η ικανότητα να συμμετέχει στην κοινωνία, υπηρεσίες ποιότητας, διότι οι υπηρεσίες πάρα πολλές φορές υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, βοηθούν τους ανθρώπους να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, αλλά και στρατηγικές απασχόλησης. Και σε περίπτωση που χάσουμε ένα από αυτά τα τρία, τότε ίσως ολόκληρη στρατηγική να καταρρεύσει. Το επόμενο κεφάλαιο και από εδώ και πέρα μπορείτε να ακολουθείτε τις ε, διαφάνειες. Θα ήθελα να σας δείξω μερικά ευρήματα σε σχετικά, σχετικά με την ανάλυση επιτυχίας που κάναμε ε, την εφαρμόσαμε σε πάνω από 25 προγράμματα σχετικά με την ενεργοποίηση της αγοράς εργασίας και και ε, συλλέξαμε, καταλήξαμε το τη συγκεκριμένη ανάλυση σε τέσσερα σημεία, σε τέσσερα γράμματα άμα θέλετε. Είναι οι προτάσεις STAR που αφορούν την συνεργασία των ενδιαφερομένων, στοχευμένες δράσεις, ε, ε, έρευνα καθώς επίσης και η υποστήριξη. Και θα ήθελα τώρα να σας πω λίγα πράγματα για κάθε έναν από αυτούς τους παραγόντες επιτυχίας θα ήθελα να ξεκινήσω με τη συνεργασία των ενδιαφερομένων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ορισμένοι από τους ομιλητές ε, δίπλα μου αναφέρθηκαν στην σημαντικότητα αυτού. Έτσι λοιπόν, άμα θέλουμε να έχουμε επιτυχημένες επεμβάσεις, ε, θα πρέπει να είναι όλοι οι παράγοντες, όλοι οι ενδιαφορέμενοι στο τραπέζι. Αρχές, ε, υπηρεσίες απασχόλησης, οι εργοδότες, ε, οργανισμοί υποστήριξη καθώς επίσης και οι ενδιαφερόμενοι άνθρωποι και οι εκπρόσωποι τους. Μονάχα αν έχουμε όλους τους παράγοντες παρόντες στο τραπέζι, στη συζήτηση, τότε μόνο θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια ιστορία, ε, μια επιτυχημένη ε, επέμβαση και νομίζω ότι είναι μια πρόκληση για αυτό το κοινοβούλιο να κατευθύνει κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε πλατφόρμες σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο, σε εθνικό, σε περιφερειακό και σε τοπικό. Όλα αυτά χρειάζονται για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε καινοτόμες στρατηγικές που θα λειτουργήσουν. Ο δεύτερος πυλώνας μιας επιτυχημένης στρατηγικής ε, είναι οι στοχευμένες δράσεις. Εντός των πολιτικών λοιπόν θα πρέπει να αναπτύξουμε στοχευμένες ε, δράσεις που θα βασίζονται σε μεμονωμένες προσεγγίσεις λαμβάνοντας υπόψη, όπως προανέφερα, τις ικανότητες των ανθρώπων. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις ικανότητες των ανθρώπων και όχι στην έλλειψη ικανοτήτων αλλά και των επιχειρήσεων, των εταιριών που δεν αναζητούν για έλλειψη ικανοτήτων αλλά για ικανότητες. Σε αυτό λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε και θα πρέπει έτσι να κάνουμε την, το, το κατάλληλο τέριασμα σε όλο αυτό σχετικά με το τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας, ένας εργοδότης. Θα πρέπει έτσι λοιπόν να εξετάσουμε ε, το, ε, την παγίδα ωφέλους ε, που είναι ένα εμπόδιο για αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα σχετικά με το πώς μπορεί να είναι μια στοχευμένη δράση. Πρόσφατα ο ΟΗΕ στην πρότασή του σχετικά με την εφαρμογή ε, της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτυγχάνει να προσλάβει ανθρώπους με αναπηρία. Έτσι λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο εδώ στις Βρυξέλλες ίσως και στο Στρασβούργο θα πρέπει να υπάρξει μια, ε, θα μπορεί να είναι μια μονάδα υποστηρικτική που θα μπορέσει να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο τρίτος πυλώνας είναι η διαθεσιμότητα υποστήριξης. Οι άνθρωποι πολύ συχνά λένε ότι ναι πρέπει να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους με αναπηρίες και ναι αυτό είναι σωστό. Όμως και ο εργοδότης χρειάζεται υποστήριξη. Το ε, νομοθετικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ πολύπλοκο ούτως ώστε να υποστηρίξει όλο αυτό. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ πολύπλοκο λοιπόν Άρα χρειάζεται υποστήριξη και για τον οργοδότη για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα αυτό τον μηχανισμό και να είμαστε σίγουροι ότι ένας, ένα άτομο με αναπηρία θα μπορέσει να εισέλθει επιτυχώς στην επιχείρηση και δεν θα είναι απλά ένα βάρος. Εμείς ως οργανισμός χαιρόμαστε ιδιαιτέρως με το πώς αυτά τα στοιχεία αυτή τη διπλή υποστήριξη περιλαμβάνονται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους ε, μακροπρόθεσμα ανέργους. Δεν παρέχει ε, υποστήριξη μονάχα στους ε, ανθρώπους με αναπηρία αλλά και στις αρχές και στους εργοδότες. Ο τελευταίο τώρα πυλώνας αφορά τις πολιτικές που βασίζονται σε έρευνα. Οι πολιτικές λοιπόν πολλές φορές βασίζονται σε ιδέες και πεπιθήσεις και όχι σε πραγματικά δεδομένα. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι πολλές φορές ανθρώπους να είναι έτοιμοι να ανακοινώσουν ότι η ανεργία σε ένα συγκεκριμένο τομέα έπεσε, αλλά αν εξετάσεις πιο προσεκτικά τα στατιστικά δεδομένα, τότε βλέπεις ότι η μακροχρόνια ανεργία αυξάνονται. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια ολιστική εικόνα και να μπορέσουμε να υποφεληθούμε τα δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί μέσω της έρευνας. Κλείνοντας λοιπόν, αυτή η ε, τριγωνική προσέγγιση είναι εντάξει, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας και τους πυλώνες και σε περίπτωση που χάσουμε έναν εξ αυτών τότε η στρατηγική ίσως να καταρρεύσει και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε ε, θετικές λέξεις πρέπει να απομακρυνθούμε από μια γλώσσα που κατηγορεί και το τέταρτο μου συμπέρασμα είναι ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει ακόμα, γι' αυτό το λόγο ας αποφύγουμε να βλάψουμε περισσότερο τις υπηρεσίες υποστήριξης όσο ακόμα υπάρχουν, να τις ε, επανισχύσουμε ξανά σε επόμενα χρόνια και έτσι να έχουμε καλά νέα. Είναι δυνατό να έχουμε ε, επιτυχημένες επεμβάσεις σε περίπτωση που εφαρμοστεί η προσέγγιση STAR. Όλα αυτά είναι που χρειαζόμαστε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζερντελού. Αναφέρατε ίσως ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσαμε να έχουμε έναν οργανισμό για άτομα με αναπηρία εδώ σε εμάς ε, στο, έχουμε δημιουργήσει το ΟΗΡΕΣ και θέλουμε ο θεσμός μας να ενισχύσει τους ετούντες εργασίας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως ένα κομμάτι του αέρας μπορεί να επικεντρωθεί στα άτομα με αναπηρία. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά τα οποία είπατε, οπότε τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Στίβεν Τόμπιν ο οποίος εργάζεται στον ε, Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, στο τμήμα χάραξης πολιτικής. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση εκ στο του Νομίζω αν σκεφτεί κανεί τους τρεις τομείς που εντοπίζονται και στη στρατηγική, αυτό που ήθελα σήμερα εγώ να συνεισφέρω στη συζήτηση είναι 10 βασικά διδάγματα που εμείς στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας θεωρούμε ότι καλύπτουν όλε αυτέ τι μέρε των τριών τομέων των δικών σα. σω ε, υπάρχει κάποια επικάλυψη όπω είπαν οι προηγούμενοι ομιλητέ, αλλά θα σα αναπτύξω τι μπορούμε να κάνουμε στο άμεσο μέλλον μετά κάποιε πολιτικέ προτάσει μέσω πρόθεσμε και ορισμένα συμπληρωματικά μέτρα με ιδιαίτερη αναφορά στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι βραχυπρόθεσμα είναι πολλά αυτά που μπορούν να γίνουν αμέσως. Το πρώτο και ίσως το πλέον σημαντικό είναι ότι οι πόροι που προβλέπονται για τι ενεργέ πολιτικέ απασχόληση να ευθυγραμμίζονται με τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε. Μεταξύ του 2011 και 2013 έχουμε δει διπλασιασμό τη μακροπρόθεσμης, ε, της μακροχρονικό διάστημα ανεργία και ακόμη και μετά συνέχισε να αυξάνεται αυτού του είδου η ανεργία με 12 εκατομμύρια άτομα παραπάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή 12 εκατομμύρια αναζητούσαν δουλειά για πάνω από ένα χρόνο. Και οι πόροι που κατευθύνονταν προς τις ενεργές πολιτικές απασχόλησης εδώ μεταξύ ε, ε, μειώνονταν και μάλιστα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πολλές χώρες ε, είχαν συρρήκνωση του ΑΕΠ τους, οπότε οι ενεργές πολιτικές απασχόλησης γνώρισαν περικοπές πιο δραστικές και από τη μείωση του ΑΕΠ. Δεν έχουμε λοιπόν ευθυγράμμιση της αντιμετώπισης με τις διαστάσεις του προβλήματος. Επίσης, από αυτή την οικονομική σκοπιά, το άλλο πρέπει να πω είναι ότι αν σχεδιάσουμε σωστά τις πολιτικές ε, της ενεργούς απασχόληση μπορεί να είναι ε, ε, ουδέτερες γιατί από οικονομικής άποψης, δηλαδή ξοδεύοντας για να βρουν οι άνθρωποι εργασία, τελικά ε, καταλήγουμε να παίρνουν κάποιο μισθό, τον οποίο όμω πληρώνουν και φόρου. Οπότε ενισχύουν τη φορολογική βάση. Δεν είναι απλώ κόστο λοιπόν, είναι μια επένδυση. Ε, επίσης, εντός του ίδια ε, συλλογιστική νομίζω είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα σενάριο που η ανεργία φτάνει το 5 και 6% αλλά μπορώ να θυμηθώ καιρούς ε, όπως τότε που εργαζόμουν στο διεθνές σκηνικό πριν από 10 περίπου χρόνια και όταν είχαμε πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας βλέπαμε συγκεκριμένες δεξιότητες να λείπουν και δώσαμε μεγάλη έμφαση, εντείναμε τις προσπάθειές μας για το πώς να επανεντάξουμε ορισμένους από όσου είναι πιο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασία. Αυτό που υπόθηκε για τη μέτρηση της απόστασης προηγουμένω. Και καταλάβαμε ότι είναι πολύ πιο δαπανηρό και πολύ πιο δύσκολο. Και παρόλο που ήμασταν σε μια φάση όπου η ενεργεία βρισκόταν γύρω στο 10%, δηλαδή τα πράγματα κάπως βελτιώνονταν σε ορισμένους τομείς, το κόστος της αδράνειας τώρα νομίζω ότι έχει γίνει πολύ μεγαλύτερο και θα αυξηθεί κι άλλο. Ε, η δεύτερη παρατήρηση για τις ε, βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις μας έχουν να κάνουν με τα ενεργά συστατικά. Τι εννοώ εδώ, η σύνθεση των ε, δαπανών και πώς γίνονται αυτές. Για να αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις δυσκολίες που υπάρχουν στο σημερινό πλαίσιο θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε θέματα όπως η κατάρτιση που δίνει υψηλή ε, επιστροφή και απόδοση σε σχέση με το βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Δηλαδή πρέπει να στοχεύσουμε τους τα μειονεκτήματα και όχι τους μειονεκτούντες απλώς. Δεν αρκεί να έχουμε ένα πρόγραμμα που απευθύνεται στους νέους. Δεν αρκεί ένα πρόγραμμα ε, για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Δεν αρκεί. Πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα ποια είναι τα εμπόδια, ποιες οι δυσκολίες τους, γιατί δεν υπάρχει συμμετοχική ε, μια αγορά εργασίας που να επιτρέπει να συμμετέχουν όλοι. Επειδή δεν έχουν δίπλωμα οδήγηση λόγω χάρη άνεργοι ή ένας άνεργος. Δεν πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε μόνο ομαδοποιημένα, πρέπει να σκεφτούμε και τα εμπόδια, τι κατηγορίε εμπόδια που αντιμετωπίζουν, δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Ε, ένα σημείο εδώ που μας ενδιαφέρει είναι ακριβώς αυτό που αναφέρω και στο 5, δηλαδή συμμετοχή ε, των κοινωνικών εταίρων και άμεση επαφή με τα άτομα. Πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν ποια είναι τα εμπόδια και δυσκολίε τους, ποιες είναι οι μελλοντικέ τους δυνατότητες και ξέρω ότι στο επίπεδο των ε, κρατικών υπηρεσιών απασχόλησης γίνεται πολλή λόγος για την τεχνολογία, τις καινοτόμες υπηρεσίες απασχόλησης. Είναι πολύ ωραία λόγια όλα αυτά, μπορεί να γίνουν και πολύ αποτελεσματικά και είναι ευπρόσδεκτη όλη η προσπάθεια. Όμω για ορισμένα από αυτά τα άτομα αυτό που χρειάζονται είναι περισσότερη επαφή, περισσότερη επικοινωνία. Και επίση σε σχέση με τη δέσμευση, την αποσύρση των κοινωνικών εταίρων. Εδώ μόνο σε συζητήσει με ομάδε μπορούμε να καταλάβουμε που είναι τα πραγματικά προβλήματα. Ε, αν ε, συζητήσουμε με κάποιον στο γραφείο μα στη Γενέβη λίγο χάρη για, τα, ε, για τις τους, ε, για το τι ε, τους λείπει, έτσι θα καταλάβουμε και θα καταλάβουν και εκείνοι τι μπορούν να κάνουν στο μέλλον και έτσι θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε την ζήτηση με την προσφορά για τις μεσοπρόθεσμες λύσεις. Για τη διαβίου μάθηση λόγω χάρη και τέτοιου είδους πρωτοβουλίες χρειάζεται επικαιροποίηση των δεξιοτήτων καθ' όλη την επαγγελματική σταδιοδρομία κάποιου. όταν κάποιος χάνει τη δουλειά του, χρειάζεται κάποια επένδυση για να επανέλθει, αλλά αν έχει διαβίου μάθηση θα είναι κάποιος που περιορισμένη επένδυση που θα χρειαστεί. Ε, Παρομοίω, αυτό που αποδίδει είναι η έγκαιρη παρέμβαση. Δηλαδή, όχι μόνο όταν κάποιος χάνει την επαφή του πρώτη φορά με την αγορά εργασίας ή με το χώρο της εργασίας, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να παρέμβουμε γέρος ακόμη και όταν κάποιος εργάζεται ή, ε, ακόμη. Ξέρω δηλαδή, σε μια δουλειά από τι προηγούμενε θέσει μου στον Καναδά, οι, οι υπηρεσίες απασχόλησης μιλούσαν με του εργοδότες, κοιτούσαν ποιοι είναι οι επικίνδυνοι τομεί και κλάδοι, πήγαιναν στο χώρο εργασία και εξηγούσαν απλώ του εργαζόμενου ότι αυτά είναι μερικά από τα προγράμματα και τι υπηρεσίε που έχουμε να προσφέρουμε αυτή τη στιγμή. Ε, έδειχναν ποια είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνταν, τα κριτήρια ρεσιμότητα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να φανούμε πιο δραστήριοι και ε, πρέπει να σκεφτούμε αυτούς που έχουν αποκλειστεί από την αγορά εργασίας με μακρόχρονικό διάστημα όμως πρέπει να σκεφτούμε αυτούς που στο άμεσο μέλλον θα χάσουν τη δουλειά τους και αυτούς που ε, μπορεί ακόμη να εργάζονται και να φροντίσουμε να υπάρξει περισσότερη δράση. Και ως προς τα συμπληρωματικά μέτρα θα επαναλάβω και εγώ ε, και μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση αυτή την ιδέα της αξιολόγησης. Και δεν εννοώ μόνο συλλογή δεδομένων με αξιολόγηση, ε, δεν εννοώ το να ορίσουμε βασικούς δείκτες, ούτε ομάδες σύγκρισης και ελέγχου, αλλά να δούμε πραγματικά τι ε, πετυχαίνει σε διαφορετικές συνθήκες. Δεν εννοούμε μόνο παρακολούθηση, ε, δεν εννοούμε ε, το 70% των ανθρώπων μπορεί να τους άρεσε ένα πρόγραμμα, 80% μπορεί να τους άρεσε ο συμβουλός τους, ούτε το 20% όσων τελικά κατάφεραν να βρουν δουλειά. Το ερώτημα είναι πόσοι, πόσοι τελικά βρήκαν δουλειά, διότι αυτό αυτό είναι η ουσία της επιτυχίας ενός προγράμματος. Εάν λοιπόν στο μέλλον δούμε τις επενδύσεις ως μέρος του σχεδιασμού ενός προγράμματος και το συνδυάσουμε με την καλή συλλογή με δεδομένων, τις καλές μεθόδους αξιολόγησης, θα είμαστε σε καλύτερη θέση και θα συζητούσαμε ίσως και σήμερα αν τα είχαμε κάνει αυτά διαφορετικά πράγματα. Βεβαίως όλα αυτά χρειάζονται και στήριξη από τις κυβερνήσεις, από τους θεσμούς, Αναφέρθηκε αυτό ήδη. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουν οι κρατικέ ε, υπηρεσίε απασχόληση, εάν θα μιλήσουν με του εργοδότε, εάν θα καταρτήσουν τεχνικέ συγκέντρωση δεδομένων, αν θα υπάρξει μια τόσα για την ε, ε, σωστή αξιολόγηση. Καταλαβαίνουμε ότι θα απαιτεί πόρου, αλλά πιστεύουμε ότι θα αποδώσει μακροπρόθεσμα πολύ περισσότερα. Και το τελευταίο που θα ήθελα να αναπτύξω και νομίζω ότι πρέπει να του δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι ναι, μπορούμε να λέμε ότι όλα αυτά είναι πολύ ωραία και σας ευχαριστούμε, αλλά τι θα γίνει αν δεν διατίθενται θέσεις εργασίας. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά τι γίνεται με τη ζήτηση. Πρέπει να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει εκεί. Ε, ε βεβαίως ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υπάρχουν εργαλεία διαθέσιμα, όπως το επενδυτικό πρόγραμμα του Juncker, το οποίο υποτίθεται ότι θα δώσει ε, όθηση στις επενδύσεις, στην ε, ζήτηση συνολικά και μάλλον θα δημιουργήσει και θέσει εργασίας. Πρόσφατα ο ILO δημοσίευσε ε, μια μελέτη για το τι επιπτώσει αναμένεται να έχει το επενδυτικό πρόγραμμα Juncker, αλλά δεν είχε ληφθεί υπόψη η συνιστόσα τη ε, απασχόληση ε, σε κάποια από τα έργα που εγκρίθηκαν και προγραμματίζονται. Όπω και δεν μπορεί αυτή η συνιστόσα να μην είναι ένα από τα κριτήρια βάσει των αξιολογούνται τα προγράμματα και τα έργα. Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν κάτι που εύκολα θα μπορούσε να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για να συνοψίσω λοιπόν, να πω ότι το μέγεθος του προβλήματος ε, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρός υπόψη και αναλόγου μεγέθους να είναι και οι λύσεις που θα προπαθούν. Θα πρέπει τα άτομα αυτά να τα εντοπίσουμε, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους τους ίδιους και τις ομάδες ανθρώπων για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, τα εμπόδια και οι δυσκολίες τους και δεν μπορούμε απλώς να στοχεύουμε ομάδες απομονωμένα αλλά να δούμε και τα ίδια τα εμπόδια, τις δυσκολίες και τις ελλείψεις. Τέλος, η διάσταση της προσφοράς και της ζήτησης θα πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει συνδυαστικά. Δηλαδή, είτε τη στιγμή που σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα, είτε εάν το σκέλος της ζήτησης ε, με μια προσέγγιση τύπου Juncker θα την ε, φέρουμε στο προσκήνιο. Και τελικώς να αναπτύξουμε και μια ανάλογη νοοτροπία υπέρ της αξιολόγησης και των ε, ε, ερευνών, των μελετών. Ω ερευνητής είναι από τα πρώτα που θα με ενδιέφερε προφανώς αυτό, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι αυτό με το πρόθεσμα μπορεί να δώσει πολύ περισσότερο ωφέλη. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστούμε πολύ. Αναφέρατε ότι το σημαντικότερο είναι να ορίσουμε τα ομπόδια. Αυτό πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό δεν πρέπει να φοβόμαστε, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να βρούμε περισσότερους ορισμούς για αυτά τα εμπόδια, για να τα γνωρίσουμε καλύτερα και να μπορέσουμε να βρούμε πώς θα τα καταρρύψουμε. Τώρα θα ήθελα να δώσω το ε, λόγο ε, τον ε, κύριο Μπέκα από το ΕΛΚ. Θα είμαι σύντομος ε, διότι άργησα να έρθω είδα το τελευταίο κομμάτι της ε, παρουσίας σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για ε, όλες τις πληροφορίες που δόθηκαν εκ μέρους σας. Ε. Δεν θα ήθελα να βγάλω ακόμα συμπεράσματα. Θα μείνω στη διαδικασία μάθησης για όταν είμαι καλύτερα προετοιμασμένος. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ από ε, τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ από την παράταξή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όλους τους ομιλητές. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μας ενημερώσατε σχετικά με την κατάσταση στα κράτη-μέλη και ότι μας δώσατε διαφορετικά παραδείγματα ενώ ταυτόχρονα αναφερθήκατε και σε θεσμούς που έχουν ένα πιο παγκόσμιο βλέμμα και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό έργο για εμάς να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι μακροχρόνια μια ανέργη και είπατε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και νομίζω Ευρώπη έχουμε ε, πολλά ακόμα να κάνουμε. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον διότι κατάγομαι από ένα κράτος ε, μέλος όπου προσπαθούμε να επανεντάξουμε τους μακροχρόνια ανέργους ε, στην αγορά εργασίας να μην τους βάλουμε απλά σε μια οποιαδήποτε θέση εργασίας ασχέτως τα κόστα απλά και μόνο για να βελτιώσουμε τις στατιστικές. Εμείς στη Γερμανία βιώσαμε αυτή την εμπειρία αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη το ότι αυτοί οι άνθρωποι γρήγορα και πάλι μένουν άνεργοι και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι το αναφέρατε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια πιστοποίηση η οποία να είναι βιώσιμη στην αγορά εργασία και αυτό απαιτεί φροντίδα καθώς επίσης και το ότι θα γίνει γρήγορα ούτω ώστε οι νέοι άνθρωποι να μην είναι άνεργοι για πολύ καιρό αλλά αντιθέτως αμέσως να μπορούν να μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Το βρήκα επίσης πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το αναφέρεται σε κάποιο σημείο, δηλαδή να αναφέρονται όλοι οι παράγοντες ε, στη συζήτηση. Όταν κοιτάω την κατάσταση στην Ισπανία έχω την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει εκεί. Στην Πολωνία τώρα βλέπω μία βελτίωση, αν το κατάλαβα σωστά μπορείτε να μου το ξαναπείτε, το γεγονός ότι ο κοινωνικός διάλογος παίζει έναν μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με πριν και το ότι έχετε επιτυχίες πάνω σε αυτό. Το δικό μου ερώτημα είναι πως ε, στην Ευρώπη έχουμε και νέες προκλήσεις όσον αφορά την αγορά εργασίας. Πώς λοιπόν πιστεύετε θα πρέπει να προχωρήσουμε διαφορετικά. Έχουμε ε, τα υπάρχοντα προβλήματα, έχουμε καλά κίνητρα, ταυτόχρονα όμως ε, έχουμε και το ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, δηλαδή να διαθέσουμε τα κονδύλια και να κάνουμε μια ανταλλαγή καλών πρακτικών, όμως κάτι τέτοιο δεν επιτυχαίνει σε όλα τα κράτη-μέλη. Έχετε κάποια συμβουλή για εμάς. Ε, μιλήσαμε για τις διασφαλίσεις για την νεολαία και όλοι εμείς Πιστεύουμε ότι αρκετά κράτη-μέλη περιορίζουν τις εγγυήσεις αυτές και με αποτέλεσμα να μην ε, ε, εξαφανίζονται ή τουλάχιστον να περιορίζονται τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν επενδύσεις σήμερα για να αποτρέψουμε μελλοντικά χρέη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα παρακαλούσα τους καλεσμένους μας να απαντήσουν πάνω σε αυτό. Θα ξεκινήσω με την κυρία Βαλέχο. Οι λύσεις πρώτα θα πρέπει να κάνουμε εκτιμήσεις με σαφείς δείκτες το τι ακριβώς γίνεται που να ξέρουμε ακριβώς σχετικά με τα ε, κονδύλια τα διάφορα και το Ταμείο Ενίσχυσης Νέων βλέπουμε ότι αποτυγχάνει καθαρά γιατί είναι ένα αποτελεσματικό το σύστημα. Δεν φτάνει τίποτα, ε, δεν φτάνει μέχρι τους νέους, δεν μπορεί να αφορά το σύνολο των νέων και τότε κανένα μέτρο δεν θα επιτύχει. Θα πρέπει να δούμε και το διάλογο με τον εργοδοτών, με τα συνδικάτα όπως επίσης και με τους νέους είπαμε, αλλά από τη στιγμή που θα μπαίνουν μόνο εμπόδια στη μέση και θα ζητάνε συνεχώς προϋποθέσεις, προϋποθέσεις, προϋποθέσεις για αυτή τη βοήθεια, τότε δεν θα γίνει τίποτα. Και αυτό σας είπα και με το πρόγραμμα δραστηριοποίησης ότι είναι μια βιτρίνα, τίποτα άλλο. Εντάξει, λένε οι Βρεξέλλες αυτό το πράγμα, το προτείνουν, το προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό, ωραίο σαν βιτρίνα, αλλά από πίσω βρίσκονται πόσες πολλές απαιτήσει, τόσα πολλά εμπόδια, ώστε δεν μπορούν να διατηθούν αυτά τα κονδύλια και να υπάρξουν μέτρα πραγματικά για να επιλύσουμε τα προβλήματα. Σίγουρα έχουμε πρόβλημα ανεργίας σίγουρα. Αλλά τι γίνεται τώρα, όλες αυτές οι περικοπές, οι συνεχείς περικοπές στην Ισπανία και εγώ σας είπα τη θέση μου με τις ε, ενεργές πολιτικές αυτές της απασχόλησης. τι γίνεται. Εδώ έθιξαν τις δυνατότητες ε, να μπορέσουν να εργαστούν κάποιοι που ήταν πρώτα άνεργοι και να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα και να μπορέσουν να ακολουθήσουν ένα δρόμο. Γιατί από τη στιγμή εσύ τους κόβεις και το προσωπικό και τις δυνατότητες και τα κονδύλια τότε τίποτα, τίποτα δεν θα πετύχουμε. Πολλά χρήματα δαπανώνται. Βέβαια θα συνεχίσουμε να ζητάμε περισσότερο αλλά τι γίνεται θα πρέπει να το κοιτάξουμε καθαρά αυτό ε, να δούμε πώς θα ξοδεύονται αυτά τα χρήματα, αλλά με τα κατάλληλα, τις κατάλληλες προϋποθέσεις, γιατί μερικές φορές τι βλέπουμε, υπάρχουν αυτόνομες περιφορίες που θα πρέπει να επιστρέφουν και χρήματα γιατί δεν τα δαπάνησαν, γιατί δεν τα χρειάστηκαν. Καταλαβαίνετε, ήταν τρομερά δύσκολες οι προϋποθέσεις οι απαιτούμενες. Ευχαριστώ. Ο κύριος καθηγητής ε, θα ήθελε να πει ίσω κάτι. Ναι, κάποια πράγματα σχετικά με τον κοινωνικό διάλογο και στο πλαίσιο της ε, πολιτικής αλλαγής ε, μετά τις εκλογές στην Πολωνία. Εγώ πιστεύω ότι ο κοινωνικός διάλογος είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό και για τη δημόσια συζήτηση. Από την έναρξη της μεταμόρφωσης η Πολωνία είχε, επέλεξε μια δύσκολη εκδοχή του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των σωματείων, των συνδικάτων και ε, των εργαζομένων. Είχαμε και την κυβέρνηση που συμμετείχε στις ε, διαπραγματεύσεις το 2013 ήταν πράγματι ένας ε, χρόνος που ο διάλογος αυτός ήταν πάρα πολύ δύσκολος για λίγο χρονικό διάστημα ε, σταμάτησε αυτός ο διάλογος και στη συνέχεια ήρθε η αποτυχία. Εγώ λοιπόν ε, συμμετείχα σε αυτόν τον διάλογο στις 11 Σεπτεμβρίου ε, υιοθετήσαμε ένα νέο νόμο που είναι άκρος καινοτομικό έδωσε την δυνατότητα να γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις και να υπάρχουν συμφωνίες όμως δεν θα ήθελα να υπερβάλλω διότι αυτός ο κοινωνικός διάλογος δεν αποφέρει πάντα καρπούς. Μερικές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως συνέβη τα τελευταία χρόνια. Είχαμε διάφορα εμπόδια όπως για παράδειγμα στο ζήτημα της ηλικίας συνταξιοζώτησης το οποίο ήταν, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και είχαμε κοινωνικές εντάσεις και έτσι δεν μπορούσαμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία όμως πιστεύω ότι παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλούμε για αυτό και άλλη μια φορά θα ήθελα όσο να, να αναφερθώ όσον αφορά τα τρία στοιχεία στα οποία αναφερθήκατε έχουμε ε, πραγματοποιήσει μια μεγαλύτερη φόρμα στην πολιτική απασχόλησή μας και στην προηγούμενη κυβέρνηση εγώ ήμουν υπεύθυνο γι' αυτό, έκανα αναλύσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να το διασφαλίσουμε, ούτω ώστε να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και θα ήθελα να σας πω το εξής. Οι δημόσιες ε, υπηρεσίες ε, εξέβρεσης ε, θέσεων εργασίας επικεντρώνεται σε αυτό. Χρειαζόμαστε επίσης όμως ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και τα λοιπά έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο διαπραγματεύσεων. Η συνεργασία είναι επίσης σημαντική ε, για μας, όπως για παράδειγμα η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από αυτήν την ε, περιθωριοποίηση, απειλούνται από αυτήν την περιθωριοποίηση, υποστηρίζονται από δύο διαφορετικές δομές από τις θέσεις εξέβρεσης εργασίας, από τα ιδρύματα εξέβρεσης εργασίας, αλλά και από ιδιωτικούς οργανισμούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους που είναι περιθωριοποιημένοι. Και η κυβέρνηση βοηθά σε αυτό και χάρη σε αυτό λοιπόν μπορούμε να δώσουμε μια εξατομικευμένη υποστήριξη και τώρα σκεφτόμαστε αν αυτές οι ικανότητες ε, στον τομέα της αποσχόλησης αν θα μπορούσαν να να ε, εφαρμοστούν για παράδειγμα να, ώστε να περιοριστεί ο ρυθμός των απολύσεων. Αντί να εισάγουμε κάτι τέτοιο θα μπορούμε να βοηθούμε τους ε, εργαζόμενους αντί να απολύουν κόσμο να αναζητούν άτομα τα οποία ίσως ε, να εκπληρώνουν καλύτερα το προφίλ που αναζητάτε. Διότι και οι απολύσεις κοστίζουν, ε, πρέπει να παρέχουμε συγκεκριμένα επιδόματα και υπηρεσίες σε αυτά τα άτομα. Κοστίζει λοιπόν. Ο εργοδότης επιπλέον θα πρέπει να συμμετέχει και στο κόστος ούτω ώστε το απολυμμένο άτομο να βρει μια νέα θέση εργασίας και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα για άλλη μια φορά να εξετάσουμε στο δημόσιο τομέα αν λειτουργεί ε, η ιδέα μας και στη συνέχεια να την εφαρμόσουμε και στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν οι τηλεπικοινωνίες ή ο, ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Εκεί γίνονται συνέχεια απολύσεις από τη μία πλευρά και από την άλλη γίνονται συνεχώς νέες προσλήψεις. Και για άλλη μια φορά το τρίτο στοιχείο τώρα, όταν ε, μιλάμε για αυτές τις ε, συνεργασίες, τις εταιρικές σχέσεις. Έχουμε την εγγυ... τις εγγυήσεις για την νεολαία, ίσως στην Πολωνία να είναι πιο εύκολο, διότι ήδη από τη δεκαετία του 90 είχαμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά από τότε, από το 95 έως το 2000, είχαμε ε, αρκετά εκατομμύρια νέους ε, ανθρώπους ε, στην αγορά εργασίας είχε αρχίσει η περίοδος αλλαγής στην Πολωνία οπότε είχαμε θέσεις εργασίας είχαμε και μια υψηλή ανεργία στο 40% και παραπάνω όμως εφαρμόσαμε αυτά τα προγράμματα για την νεολαία και μάλιστα πριν γίνουμε κράτος μέλος της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε τέτοια ε, προγράμματα, είχαμε δηλαδή προετοιμαστεί για αυτές τις εγγυήσεις. Άρα εκτός από αυτό που κάνουν ε, οι υπηρεσίες απασχόλησης και σε περιφερειακό επίπεδο έχουμε κάποια προγράμματα αλλά έχουμε και ένα διαφορετικό μοντέλο όπως ε, για παράδειγμα μια ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα. Κάποιος ο οποίος δηλαδή γράφει τη διπλωματική του εργασία, ένας φοιτητής ε, με τον επιβλέποντα της διπλωματικής του μπορεί να ξεκινήσει ένα κοινό πρόγραμμα για παράδειγμα, το οποίο θα λάβει μια κάποια χρηματοδότηση και θα έχει ε, θα οδήγησε σε 3.900 νέες startups. Συγγνώμη που μίλησα τόσο πολύ. Σβέν, θα ήθελες να πεις κάτι. Πολύ σύντομα. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούστηκαν είναι γιατί δεν προτείνονται νέε λύσει. Με έχουν αποσχολήσει τα προγράμματα απασχόληση επί μακρόχρονικό διάστημα. Είναι πολύ δύσκολο να βρει κανεί μια ιδέα ρηξικέλευτη, διότι Συνήθως αυτό που χρειάζεται είναι ότι κάποιος θέλει κάποιες δεξιότητες παραπάνω, επαφές με εργοδότες, κάτι τελείως καινούριο είναι λίγο δύσκολο. Το να συνδυαστούν με νέο τρόπο ε, κάποιες γνωστές ιδέες, το να καταλάβει κανείς ότι υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στην ίδια διαδικασία, αυτό ναι. Ένα παράδειγμα που προέκυψε αρκετές φορές στη συζήτηση, αλλά να το δώσω ίσως έμφαση. Νομίζω στις Ενεργέ πολιτικέ. Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στο τι γίνεται τη στιγμή που καθώ χάνει τη δουλειά του. Αυτό που παραβλέπουμε είναι κάποια πράγματα που μπορούσαν να έχουν γίνει από πριν για να αποφύγει κανεί την ανεργία. Δηλαδή, ενώ εργάζεται, τι μπορεί να του προσφέρουμε, πώ να τον στηρίξουμε για να μείνει στη θέση εργασία του. Καλύτερε συνθήκε απασχόληση και μια καλύτερη σταδιοδρομία μπροστά του. Ένα-δυο παραδείγματα. Για την πρόληψη. Είναι πολλές οι χώρες που έχουν ε, δει ότι αυτοί που έχουν τα τελευταία χρόνια επίδομα ενεργείας, το 1 τρίτο τουλάχιστον, είναι άνθρωποι με ναι, ενήλικες μάλλον, με κάποια προβλήματα ε, ψυχολογικά. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για τους ανθρώπους αυτούς πριν ε, χάσουν τη δουλειά τους, πριν βρεθούν στο χώρο της ενεργείας. Υπάρχει ένα κοινωνικό στίγμα στην κοινωνία μας. Εάν έχει κανείς ε, προβλήματα υγείας και ζητήσει βοήθεια ή αν ε, ένας δάσκαλος φανεί ε, στους μαθητές ότι έχει πρόβλημα, κάποιες συναισθηματικές διαταραχές, αυτά όλα δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να εκπαιδεύσουμε δασκάλους, εργοδότες, τους συμβούλους της Δημόσιας Απασχόλησης, στους γιατρούς, τους παθολόγους που εντοπίζουν στην αρχή αυτά τα προβλήματα συνήθως να τους δώσουμε ιδέες για το πώς να ε, ευαισθητοποιήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Να αρχίσουν να μιλάνε για το πρόβλημα και να προτείνουν λύσεις όταν εντοπιστεί. Αλλά και φορείς ώστε, το πρόβλημα, όταν εντοπιστεί το πρόβλημα να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει βοήθεια ειδικού. Κάποιοι που είναι επιμακρών ε, άνεργοι μπορεί να χρειαστούν επί μεγάλο χρονικό διάστημα υποστηρικτική παρουσία για να περάσουν στην αγορά εργασίας και αφού ξεπεράσουν την ανεργία. Έτσι λοιπόν να επικεντρωθούμε στο, όχι μόνο στο χρονικό σήμα που κάποιο χάνει τη δουλειά του, αλλά και στο τι έρχεται πριν και μετά. Ευχαριστώ. Απλώς λίγα λόγια, λίγα γενικά σχόλια Πρώτα απ' όλα για τον κοινωνικό διάλογο. Βεβαίως ο κοινωνικός διάλογος είναι απολύτως αναγκαίος, ζωτική σημασία εργοδότες και εργοζόμενοι, αλλά και επίσημοι φορείς να καθίσουν και να συζητήσουν όταν σχεδιάζουμε αυτές τις πολιτικές, αλλά δεν αρκεί αυτό, δεν φτάνει. Πρέπει να συμπληρωθεί και από τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και αυτοί θα πρέπει να πάρουν μέρος στις συζητήσεις. Το είπα στο πρώτον πυλώνα για τι. Ε, επιτυχημένες ενεργές ε, στρατηγικές. Επίσης πρέπει και οι ίδιοι οι να εκπροσωπούνται στις συζητήσεις. Ιδάλλως μπορεί κάτι να χαθεί, να παραλυφθεί και να μην έχουμε την ανάλογη αντιμετώπιση που χρειάζεται για την κάθε ομάδα. Σε ό,τι αφορά τις νέες προκλήσεις στην αγορά εργασίας και πώς αντιμετωπίζονται. Ο δικός μου οργανισμός συγκέντρωσε ήδη δύο φορές ε, κάποια πρότυπα καλών πρακτικών κάποια μοντέλα που τα έχουμε μελετήσει και έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν στον τόπο μας σε διαφορετικές γλώσσες και ήδη έχουμε απονείμει μετάλλιο, παράσιμο σε κάποιους από τους οργανισμούς που τα πήγαν ιδιαίτερα καλά. Έχουν αναπτύξει μεθόδους προσεγγίσεις που έχουν δώσει αποτελέσματα. Μία από τις μεθόδους που ε, έχει αποδεχθεί επιτυχημένη είναι οι εργοδότες να καλλιεργήσουν την ε, πολυμορφία στο χώρο εργασίας. Το έχουμε συζητήσει με ερευνητές και το επιβεβαιώνουν μελέτες ότι η διαφοροποιημένη, η ποικιλόμορφη ε, εργατική δύναμη εργάζεται καλύτερα. αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να το γνωρίζουν και οι εργοδότες και να το καλλιεργούν. Και αυτό που κάναμε επίσης με τα υψηλότερα στελέχη του management κάποιων εταιριών είναι αυτό που ονομάζουμε η, ο σχεδιασμός μιας θέσης εργασίας. Δηλαδή κοιτάζουμε ένα άτομο και τι δεξιότητες έχει, τι μπορεί να προσφέρει και κοιτάζουμε πώς θα τον ε, ε, τοποθετήσουμε σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις εργασίας που μπορεί να ταιριάζουν με αυτές τις ικανότητές του. Έτσι είναι ευκολότερο να βρει κανείς αξιοπρεπείς θέσεις με καλές, με, καλέ, με αμοιβές και για ανθρώπους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή με αναπηρίες. Έτσι μπορούμε να καταρτήσουμε καλύτερες στρατηγικές πιο επιτυχημένε. Ω προ την εγγύηση για του νέου, αναφέρθηκε πολλέ φορέ. Στι περισσότερε χώρε αυτό εφαρμόζεται ω ένα εξάμεινο εγγύηση Υπόθηκε προηγουμένως για ανθρώπους με ε, κάποιες αναπηρίες, με ψυχοκοινωνικά προβλήματα όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Έξι μήνες δεν φτάνουν. Πρέπει να υπάρχει διαρκής στήριξη ε, και πρέπει να καθορίσει κανείς ε, μια ολόκληρη πορεία για τη σταδιοδρομία του εφόσον θέλει να είναι επιτυχημένος στις παρεμβάσεις του. Ε, πέρα λοιπόν του κοινωνικού διαλόγου, η εμπλεκόμενοι σε αυτές τις συζητήσει πρέπει να χρησιμοποιήσουν και νοτόμα πρότυπα και ε, μια πορεία για την ε, καριέρα, για την επαγγελματική σταδιοδρομία που είναι πολύ σημαντική, ώστε όχι απλώ να φέρουμε πίσω του ανθρώπου στο χώρο εργασία, αλλά και να του κρατήσουμε εκεί. Και τελευταία παρατήρηση, δεν αναφέρθηκε μάλλον ακόμη σήμερα εδώ, κάτι που πρέπει να κοιτάξουμε είναι ε, όλο ο μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο προσφέρει μεθόδου για να είμαστε ακόμη πιο συνεκτικοί στην αντιμετώπιση μα. Να επιδιώξουμε ακόμη επιτυχέστερα του τρόπου που συζητάμε, του στόχου που συζητάμε εδώ. Η αγορά εργασία είναι ένα θέμα πολύ περίπλοκο, διάστατο και πρέπει να το δούμε αυτό με έναν τρόπο συντονισμένο. Πρέπει ιδέες ώστε οι ιδέες που ακούσαμε από τους διάφορους ομιλητές ε, σήμερα να μας οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τόμπιν. Θέλετε να απαντήσετε. Θα περιοριστώ τα σχόλια μου ε, στην μακροχρόνια ανεργία που θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Αρχικά τι μπορούμε να κάνουμε για τους μακροχρόνια ανέργους Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για τα μέτρα, τις ε, πολιτικές ε, και όλα αυτά είναι ωραία και καλά. Νομίζω ότι όσον αφορά τους μακροχρόνια ανέργους ε, το ζήτημα, υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα, το γεγονός ότι τα ποσοστά είναι υψηλά σε μερικές περιπτώσεις όμως αυτό δεν είναι παντελώς κακό. Είναι κακό το γεγονός ότι 12 εκατομμύρια άνθρωποι ψάχνουν πάνω από ένα χρόνο για να βρουν δουλειά. Όμως είναι καλό πράγμα το ότι ξέρουμε πως ακόμα ψάχνουν για δουλειά. Σε παλαιότερες κρίσεις αυτό που έχουμε δει οι μακροχρόνια άνεργοι μειώνονται εις βάρος των ανθρώπων που τα παρατούν εντελώς. Τι μπορεί, λοιπόν να, τι, τι μπορεί λοιπόν να γίνει τώρα για, την, για τους μακροχρόνια ανέργους είναι να διασφαλίσουμε ότι έχουν πρόσβαση στα υπάρχοντα προγράμματα υποστήριξης ε, Κάποιοι θα χάσουν τα επιδόματά τους, ίσως θα χάσουν ε, τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κάποια προγράμματα εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτοί οι 12 εκατομμύρια άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα, σε όσο το μεγαλύτερο βαθμό αυτό είναι δυνατό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα ε, να καλέσω και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ε, να συμμετάσχουν ε, στη συζήτηση. Αρχικά ο κ. Πυρίντσκι θα σας παρακαλούσα να περιοριστείτε σε δύο λεπτά παρακαλώ. Αν πιστεύετε ότι θέλετε να απευθύνετε ένα ερώτημα σε κάποιον συγκεκριμένο, τότε μπορείτε να το κάνετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σίγουρα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, πέντε παρουσιαστές ε, για ε, τις ερευνές τους, τις παρουσιάσεις τους. Ένα ερώτημα θα ήθελα όμως να θέσω και αυτό αφορά, με, αφορά τον κοινωνικό διάλογο. Εμείς οι σοσιαλιστές δίνουμε ιδιαίτερο βάρος ε, στην ε, κοινωνική ε, συνεργασία και εγώ θα ήθελα να το ονομάσω αυτό καλύτερα συλλογικές διαπραγματεύσεις διότι η ενεργό συμμετοχή σημαίνει συμμετοχική αγορά εργασία, θέση εργασίας μαζί με επαρκή κοινωνική προστασία και αν επιστρέψουμε στο πρώτο ε, ζήτημα της υποστήριξης επαρκούς εισοδήματο, ε, το οποίο αναφέρατε μερικοί από εσά, είναι μια δουλειά που πληρώνει ουσιαστικά. Και μία άλλη ανησυχία για αυτό το θέμα που μοιραζόμαστε είναι ότι δεν μπορούμε να μιλούμε για θέσεις εργασίας και απασχόληση, αλλά για θέσεις εργασίας ποιότητας. Δουλειές οι οποίες έχουν νόημα και όπως λέτε εσείς ε, ε, παρέχουν δυνατότητες ε, καριέρας, ανάπτυξης και βγάζουν μπροστά τις ε, ικανότητες του εργαζόμενου. Νομίζω λοιπόν ότι αξίζει να εξετάσουμε τις εμπειρίες και να βγάλουμε τα πασιφανή συμπεράσματα ε, για χώρες που εφαρμόζουν συλλογικές διαπραγματεύσεις ε, και προωθούν μια ε, κοινωνική οικονομία. Κάποιος μπορεί να σκέφτεται το αναρχικό μοντέλο ή κάποια μοντέλα της κεντρικής Ευρώπης. Εκεί η κατάσταση είναι κάτω από το μέσο όρο και γενικότερα η ποιότητα θέσεων εργασίας συμπορεύεται με μια δέσμευση ε, κοινωνικής ε, εταιρικής ευθύνης όταν λοιπόν συζητούμε για, ενεργές, ε, για πολιτικές ενεργής αγοράς, της αγοράς εργασίας πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποια σημεία κλειδιά τα οποία κάνουν την διαφορά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους ε, καλεσμένους ε, για τις παρουσιάσεις τους. Εμείς εδώ πάρα πολύ συχνά ε, δημιουργούμε προγράμματα τα οποία σχηματίζουν ένα πλαίσιο, όμως δεν εξετάζουμε πώς εφαρμόζονται νομοθετικά και εδώ σκέφτομαι την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ατζέντα για νέες ικανότητες, ε, την πρωτοβουλία ε, κινητικότητας των νέων, πρωτοβουλίες ε, για τις οποίες έχουμε εργαστεί πάρα πολύ, αλλά και οι εγγυήσει για την νεολαία εδώ και, πάνω από, εδώ και μήνες ασχολούμαστε με αυτό και γι' αυτό το λόγο με εκπλήσει λιγάκι όταν ακούω ότι σε διάφορα κράτη-μέλη αξιολογείται ως αποτυχία, όπως είναι για παράδειγμα στην Ισπανία. Αυτό με εξέπληξε. Όμως γνωρίζω ότι τα κράτη-μέλη πολύ συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες να δημιουργήσουν ε, προγράμματα ε, στα οποία ελάχιστα κράτη-μέλη έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οπότε υπάρχει μια τεράστια ανισότητα, ανισότητα κατά τη γνώμη μου και όσον αφορά τα διάφορα σχολικά συστήματα. Μιλάμε συνεχώς για διαβίου μάθηση. Όμως η βάση, τα σχολικά συστήματα, από εμπειρία το λέω, ξέρω ότι διαφέρουν πάρα πολύ και απέχουν πάρα πολύ από το να ε, κοιτούν προς την αγορά εργασίας. Και δεν γνωρίζω μια λύση για αυτό, όμως ε, στη γενικότερη συζήτηση θα μπορούσε να προκύψει κάτι εκεί. Όσον αφορά τις, ε, τους οργανισμούς εργατικού δυναμικού. Και εκεί, κυρίες και κύριοι, λέτε ότι θα πρέπει να έχουν τους αναγκαίους πόρους, τη γνώση αλλά και τους πόρους, ούτως ώστε να μπορούν να παρέχουν κάποια βοήθεια. Λέτε ότι δικαίως ότι κάθε ε, περιστατικό είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και χρειάζεται η αντίστοιχη βοήθεια, όμως συνειδητοποιώ ότι οι οργανισμοί αυτοί δεν είναι ιδανικοί γιατί δεν έχουν καν τη δυνατότητα, οπότε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι και εγώ... Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ειδικού οι οποίοι ήρθαν σήμερα το απόγευμα εδώ και οι οποίοι έκαναν τις εισηγήσεις τους πραγματικά ωφέλιμες. Θα ήθελα να σας πω ότι σχετικά με την προσαρμογή στην αγορά εργασίας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μας. Ίσως ο κ. Μεντσίνα δεν το είπε ανοιχτά, αλλά για την Πολωνία ήταν κάτι το πολύ σημαντικό γιατί επήλθε μια σημαντική αλλαγή σχετικά με τη χρηματοδότηση για τη, ε, για, από πλευράς δημοσίου. Και στο παρελθόν, παλιότερα, υπήρχε χρηματοδότηση ακριβώς για μια κατάρτιση, ενώ τώρα τα κέντρα αυτά παίρνουν τα κονδύλια μόνο εάν μπορέσουν τελικά να ενταχθούν στην αγορά εργασίας οι εργαζόμενοι ή να διατηρήσουν ε, την εργασία τους. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματικότητα και προσαρμογή στην αγορά εργασίας. Διαφορετικά Χωρίς κάτι τέτοιο τότε ο άνεργος δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να πετύχει την ανταξή του. Με την αλλαγή αυτή είχαμε και πολλές νέες δραστηριότητες από πλευράς των κέντρων αυτών για την απασχόληση. Και γι' αυτό χρειάστηκαν και οι εταιρικές σχέσεις, συνεργασίες για τις οποίες μιλήσαμε προηγμένως. Συνεργασίες με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με εργοδότες κλπ. Μερικές φορές ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι ακριβώς εξειδικευμένες ε, για να ευνοήσουν και άτομα με αναπηρίες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε και για την εκπαίδευση, για κατάρτιση σε κατάλληλα κέντρο, κέντρα, το προσωπικό θα πρέπει να μπορεί να συνεργάζεται αυτό που εργάζεται εκεί. Το προσωπικό να έχει τις απαραίτητες δεξιότητες, τα προσόντα για να βλέπει ποιος είναι ικανός γιατί από όσους απευθύνονται στα κέντρα αυτά. Και τα προσόντα αυτά σίγουρα είναι δύσκολα να τα αποκτήσει κανείς, αλλά κάποιος θα πρέπει να τα διδάξει. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να τα διδαχθούν. Η προσαρμογή στην αγοραγασία είναι πολύ σημαντική και υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι για να την πετύχει κανείς και ακόμα μιλήσαμε για μία πρόκληση. Για μία πρόκληση που είχε να κάνει για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες για την προσαρμογή στην αγορά εργασίας. Έχουμε τρεις κύριες προκλήσεις. Πρώτα απ' όλα τη δημογραφική πρόκληση. Ε, παρατηρείται γύρανση του πληθυσμού. Δεύτερη πρόκληση είναι η ψηφιοποίηση, σχετικά με την πληροφορική δηλαδή κλπ της αγοράς εργασίας και καταλαβαίνετε ότι όσοι έχουν μια κάποια ηλικία αποκλείονται από την αγορά εργασίας επειδή δεν έχουν γνώσεις πώς ε, θα ασχοληθούν με τους υπολογιστές. Και αυτό αφορά οποιοδήποτε εργαζόμενο, οπουδήποτε από τη στιγμή που μπήκε στη νέα εποχή της πληροφορικής η εταιρεία του που χρειάζονται ειδικά προσόντα, απαραίτητα. Λοιπόν, όταν μιλάμε για αποτυχίες, το πώς δεν καταφέρνουν πάνω από 50 ετών τους εργαζόμενους να τις επανεντάξουν, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το φαινόμενο αυτό τις ε, ανάγκες που υπάρχουν για γνώσεις πληροφορικής. Το τρίτο και τελευταίο που περιορίζει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ποιο είναι ότι διαφέρει από εθνικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής πλευράς η Ευρώπη στις διάφορες περιοχές της. Και αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε, δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Ήδη είναι εντελώς διαφοροποιημένη η κοινωνία, τη μια μεριά στην άλλη, και αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν είμαστε σε θέση να πετύχουμε ώστε αυτή η διαφορετικότητα να την υπόψη και από τους εργοδότες. Στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη κυρίως αυτή η πτυχή είναι, αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση. Αν θέλουμε να έχουμε μια πολιτική ισότητα στην αεροργασία θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο κάθε εργαζόμενος είναι διαφορετικός από τον διπλανό του και τον παραδιπλανό του. Υπάρχουν πολλοί με υψηλές δεξιότητες, αλλά Ίσως δεν χρειάζονται μερικές θέσεις αυτά τα υψηλά προσόντα. Η κατάσταση επιδεινώνεται στην Ευρώπη. Όσοι εσείς εκπροσωπείτε, το καταλαβαίνουν ότι αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες αυτούς το μισθή, όχι. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Βαλέχο Μιλήσατε για τις εγγυήσεις νεολαίας στην Ισπανία και είπατε ότι ήταν ένα φιάσκο οφείλεται στο γεγονός ότι αρχικά τα κράτη-μέλη, υπήρχαν κράτη-μέλη τα οποία δεν είχαν οικονομικά μέσα για να αρχίσουν αυτό το πρόγραμμα και γι' αυτό το λόγο ήταν αποτυχία. Και το δεύτερο ερώτημα, υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Είχατε μεγάλες επιτυχίες όσον αφορά ε, τα εργατικά σωματεία. Μπορείτε λοιπόν να το φέρετε αυτό σε επαφή με τα σωματεία. Και έχω και ένα ερώτημα για τον κύριο Μετσίνα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όταν οι καταρτήσεις χρηματοδοτούνται κατά 100% ε, αυτό είναι μια καλή λύση ε, ή όχι. Μήπως θα έπρεπε και οι εργοδότες να συμμετάσχουν ε, με τη χρηματοδότηση διότι ίσως έτσι να σέβονται καλύτερα τους εργαζομένους τους, ε, ίσως να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι έτσι. Και ένα ακόμα ερώτημα. Ε, μας γνωστοποιήσατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε ότι άνθρωποι που δεν έχουν κίνητρο ή αποτελούν μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Ο κύριος Βάιμ είπε πόσο, πόσο σημαντικό είναι το να υπάρχουν κίνητρα τι μπορούν να κάνουν λοιπόν οι επιχειρήσει, ούτω ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν κάποιο κίνητρο να επιστρέψουν στην αγορά εργασία. Και τρίτον, έχω ένα ερώτημα για τον κύριο Πολ Σουέιμ σχετικά με τα κίνητρα μιλήσατε θετικά για το θέμα αυτό και είπατε πόσο, είναι, πόσο, απε, σημαντικό είναι να υπάρχει κίνητρο και η κοινωνία ανεξαρτήτως ηλικίας να μην περιθωριοποιεί κάποιες ομάδες. Μερικές φορές μάλιστα δεν γνωρίζουμε καν ότι κάποια ομάδα μέσα στην κοινωνία έχει περιθωριοποιηθεί πολλές φορές ε, πρόκειται για ομάδες αξιόλογων ανθρώπων, πολύτιμων ανθρώπων. Και ένα ακόμα ερώτημα προς τον ε, κύριο Λουκ Ζελντερλού. Είπατε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Είπατε ότι ο εργοδότης θα πρέπει ε, να εκμεταλλεύεται μια θέση εργασίας και τη συγκεκριμένη ιδέα την βρήκα πάρα πολύ καλή. Όλοι μας έχουμε εργαστεί σε κάποια ομάδα, όλοι μας σκεφτόμασταν ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε τη δουλειά στα μέλη της ομάδας και έτσι λοιπόν το ερώτημά μου είναι τι πρέπει να κάνουμε ούτω ώστε οι εργοδότες να κατανοήσουν αυτή τη φιλοσοφία για να καταλάβουν ότι ότι ε, μπορούν να προσαρμόσουν τη θέση, εργασ... τη, θέση... τη θέση εργασίας στους εργαζόμενους. Και ένα ερώτημα για τον κύριο Τόμπιν. Ε, αναφερθήκατε στις εμπειρίες σας από τον Καναδά και ότι οι Καναδοί κινητούν μακριά στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι δύσκολο τώρα να πούμε ε, ε, ποια επαγγέλματα θα χρειαζόμαστε σε 2, 5, 10 χρόνια. Όμως εμείς στην Πολωνία είχαμε κάποτε τέτοια προγράμματα. Είχαμε προγράμματα με τους Γερμανούς αλλά και με ανθρώπους από τη Δανία. Και στην δική μου περιοχή κάθε κοινότητα ήταν υποχρεωμένη να συλλέξει 100 εργοδότες και να τους ρωτήσει ποιους θέλετε να απολύσετε, ποιος θέλετε να επαναπροσλάβετε και τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αλλά στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε και το ξεχάσαμε. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να επιστρέψουμε σε τέτοια προγράμματα. Νομίζω ότι θα, κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ πολύτιμο. Και είπατε και κάτι ακόμα. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να εξαλείψουμε τα προβλήματα ε, στην απασχόληση. Ε, είπατε πόσο σημαντική είναι η κατάρτιση, η εκπαίδευση. Το σχολείο σήμερα οι άνθρωποι χρειαζόνται εκπαίδευση, άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου ικανότητες. Όμως τέτοιες ικανότητες όπως η στρατηγική σκέψη ή η ικανότητα λήψης αποφάσεων. Όλα αυτά θα πρέπει να ξεκινούν από τον υπηαγωγείο, με παιχνίδια για παράδειγμα. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν αυτές τις ικανότητες και στη συνέχεια δεν χρειάζονται περαιτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα για να αποκτήσουν τις συγκεκριμένες ικανότητες όταν μεγαλώσουν. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να απαντήσετε τα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω σε ερωτήσεις ε, και στον πρώτο ομιλητή. Γι' αυτό το Ταμείο Ενίσχυσης των Νέων ε, Εγγύησης ε, για τρία χρόνια ακούσαμε πολλά και διάφορα να λέγονται και λίγα είδαμε να γίνονται. Ότι εντάξει τώρα θα λύναμε τα προβλήματα των νέων μας αλλά τη στιγμή που έπρεπε να λειτουργήσει δεν μας έδινε καρπούς. Τίποτα. Εντάξει, διάφορα εργαλεία και τα λοιπά είπαν ότι ας πούμε θα έπρεπε οι νέοι να είναι εγγεγραμμένοι σε καταλόγους ώστε οι αυτόνομες περιφέρειες να συντάξουν προγράμματα και λοιπά, να βλέπαν ποιος έχει τι και λοιπά και να δούνε τι γίνεται ανάλογα με την ε, με, την, ε, με τις ρυθμίσεις. Από λεωφορικής πλευράς ήταν ε, καταστροφικό αυτό, καταλαβαίνετε. Μπερδευόταν όλοι. Υπήρχε κόσμος που ήταν γεγραμμένος κλπ. Αλλά εκεί οι απαιτήσει όπως βέβαιναν αυτά ήταν τόσο μπερδεμένα και δεν έδωσαν τίποτα, κανένα θετικό αποτέλεσμα στους νέους μας. Και ήταν φιάσκο, αποτυχία και εντάξει έγινε προσπάθεια να κινηθούν διάφορα προγράμματα από λεβάς κεντρική κυβέρνηση. Όμω δεν έδιναν χρήματα, κονδύλια. Και αυτό το συνδυάζω με την πρώτη μου παρέμβαση που είπα ότι έκανε περικοπές το 66% των ενεργών πολιτικών ε, ε, απασχόλησης η κεντρική κυβέρνηση. Γι' αυτό ακριβώς δεν είχαν τα κονδύλια στη διάθεσή τους οι περιφερειακές κυβερνήσεις ε, για να μπορέσουν να προχωρήσουν να περπατήσουν προγράμματα για να μπορέσουν να ενισχύσουν τους νέους με τις καταλαβαίνετε ταμείο κλπ. Καταλαβαίνετε με αυτές τις περικοπές. Αυτές οι περικοπές ήταν και περικοπή πολιτικών, αποτελεσματικών και δραστηρίων και ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκαν κυνηγώντα, τρέχοντας πίσω, τιμωρώντας αυτούς που προσπαθούσαν ε, γιατί και κονδύλια πήγαιναν ε, αλλού και όχι εκεί στα οποία, στους στόχους που προοριζόταν από την αρχή, όχι για την απασχόληση. Γιατί υπάρχουν τα χρήματα για να γίνουν αυτά και όχι αντίθετα από ό,τι λέει, λένε οι Βρυξέλλες. Είναι τελικά υπέρ των περιοχών που δεν έχουν τόσες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, Εκεί θα, αυτές θα πρέπει να ενισχυθούν και όχι οι πλουσιότερες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν. Εδώ έχουμε ένα ικανό ποσοστό κατά το οποίο μειώθηκε η ενίσχυση αυτή και τελικά ορισμένε περιφέρειες έχουν χρήματα, άλλε όχι. Θα μπορέσουν λοιπόν, πρέπει αυτές οι περιφέρειες να μπορέσουν να αναπτύξουν τα προγραμμάτά τους. Εκείνες που δεν είχαν χρήματα δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και ήταν εκείνες που υπέφεραν και περισσότερο. Και τώρα λέει εντάξει κάποιος άνεργος, νέος άνεργος, αλλά λησμονούν ποιες πολιτικές θα πρέπει να ασκηθούν για να λύσουμε τα προβλήματα αυτών των νέων. Η πρώτη ερώτηση, η πρώτη παρέμβαση που είχε να κάνει με τον κοινωνικό διάλογο και την συλλογική διαπραγμάτευση αυτά τα δύο έπρεπε να εξεταστούν και πρακτικά αυτή η περιγραφή πριν από αυτά που είπα εγώ μέχρι το Μάιο του 2015. Οι ήταν διάφορες περιοχές στην Ισπανία γιατί δεν υπήρχε κοινωνική διαπραγμάτευση και για να γίνει κάτι τέτοιο εκεί που γινόταν όμως δεν εφάρμοζαν αυτά που συμφωνούσαν κατά τη διάρκεια του κοινωνικού διαλόγου. Τι έγινε και αναφέρομαι στην Καστιλιά Λαμάντσα, γιατί εκεί ξερίζωσαν κάθε σωστή πολιτική, απολύτως όλες τις σωστές, έτσι, ναι, εκ των πραγμάτων. Και ξέρετε που φτάσαμε, ότι επιστράφηκαν κονδύλια χρήματα επειδή δεν τα διάθεσαν, καταλαβαίνετε. Ε, αυτά, έτσι έχει υπόθεση. Τώρα τι έγινε αυτά τα τέσσερα χρόνια τα συνδικάτα. Το Κομισιόν Σομπρέρα, το δικό μου το συνδικάτο, είπε ότι χρειαζόταν η προστασία αυτών των ατόμων. Ε, γιατί αποτελούσε αδικία αυτό που συνέβαινε. Ε, έπρεπε στην ε, αγορά εργασίας να μπορούσαν να ενταχθούν και μάλιστα ποιοτικά. Το Μάιο η νέα κυβέρνηση συναντήθηκε με τους εργοδότες και τα συνδικάτα και μαζί με τα συνδικάτα και την πρότασή μας ξεκίνησε και έληξε προθεσμία μία εβδομάδα πριν, ξεκίνησε μία πρωτοβουλία από πλευρά του Συνδικάτου Κομισιόνε Σομπρέρας τα εργατικά, εργατικές επιτροπές, ακριβώς ε, για διάφορα χρήματα ε, για κόσμο, κονδύλια για κόσμο που δεν έχουν κανένα εισόδημα και να μπορέσει να υπάρξει ένα συμβόλαιο πλήρους εργασίας επί έξι μήνες ε, σήμερα και με τη συλλογική σύμβαση ώστε έτσι μετά από τους έξι μήνες να δουν πώς να μπορέσουν να συνεχίσουν να προστατεύονται κοινωνικά ε, και από την ανεργία μέχρι και 21 μήνες θα μπορούσαν να προστατευτούν με κάποια ενίσχυση, ακριβώς άτομα που είχαν οικογένεια, παιδιά κλπ. Και εμείς διαπραγματευτήκαμε και τον Νοέμβριο και λέγαμε ότι ήταν ανοησία του ισπανικού συστήματος αυτά τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια ότι διαλύθηκε η δημόσια υπηρεσία που ασχολιόταν την, με την απασχόληση και θα έπρεπε μαζί με τα συνδικάτα μια συμφωνία και με την κυβέρνηση με αυτά τα τελευταία που έγιναν για να μπορέσει να υπάρξει μια διαπραγμάτευση, να δοθούν κονδύλια για τουλάχιστον 80 άτομα που θα προσληφθούν τώρα σε, αυτά τα, σε, αυτές τις υπηρεσίες του δημοσίου για να ασχοληθούν με την ένταξη. Να πρέπει να δούμε μετά την ε, κοινωνικό διάλογο ή μη κοινωνικό διάλογο, να δούμε τι έχει γίνει. Και στην Καστήλια Λαμάντσα, σε αυτά αναφέρομαι, γιατί και εδώ παρακαλώ, παρακαλώ πώς μπορείτε να ολοκληρώσετε, λέει πρόεδρος, γιατί περνάει η ώρα και θα πρέπει να μιλήσουν όλοι. Ναι, ναι, οι πολιτικές απασχόλησεις που ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα και μας ζήτησαν μαζί με τη συνδικάτα και τους εργοδότες να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 duży problem jak gdyby po Ευχαριστούμε ο Σουέιμ. Ευχαριστώ. Αυτό που μόλις είπε ο τελευταίος ομιλητής για τα κίνητα και την κινητοποίηση είναι ακριβώς το σωστό. Ε, η ερώτηση αλλά και το φως που ρίξατε στην όλη υπόθεση ήταν πολύ εύστοχο. Είναι απλό να κοιτάζουμε ποιοι έχουν δυσκολίες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να κρίνουμε αν έχουν αρκετά κίνητρα ή όχι. Αλλά το θέμα είναι το κατά πόσον εμεί κατανοούμε τι δεξιότητέ του και το κατά πόσον έχουμε σωστή επικοινωνία μεταξύ του. Υπάρχει λοιπόν μια σχέση διαδραστική, δυναμικού χαρακτήρα. και για τους ανθρώπους με αναπηρίες και για τους ενδεχόμενους εργοδότες λοιπόν αλλά και τους εργαζομένους της υπηρεσίας απασχόλησης των κρατών πρέπει να δούμε τι μπορούμε να τους προσφέρουμε. Οι περιθωριοποιημένες ομάδες στην κοινωνία πρέπει να ε, έχουν επίγνωση. Ε, ένας από τους προηγούμενους ομιλητές μίλησε για τι μελλοντικέ προκλήσει στην αγορά εργασία, όπω ο κύριο του πληθυσμού. Αυτέ τι ομάδε έχουμε σκεφτεί. Πρέπει να ξαναδούμε ποιοι είναι οι ενδεχόμενοι ρόλοι των ηλικιωμένων στην αγορά εργασία πώς μπορεί να εκμεταλλευτούμε το χρόνο που θα διαθέτουν υπέρ μας. Πρέπει λοιπόν να δούμε και την μεταβολή της, του πληθυσμού των εργαζομένων, το κατά πόσον γυράσκει όχι και τι ε, επιπτώσεις θα έχει αυτό το φαινόμενο. Ε, πάντως, υπόθηκε ότι υπάρχουν πολλές ε, αλλαγές στην αγορά εργασίας ε, πρέπει να το δούμε και από τη σκοπιά του κοινωνικού διαλόγου, διότι η ψηφιοποίηση, η γύρα του πληθυσμού, η, η πολυμορφία είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους τους κοινωνικούς εταίρους στην, θα έπρεπε να ενδιαφέρει όλους τους κοινωνικούς εταίρους στην κοινωνία και να μπορεί να ακουστεί η φωνή τους. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λουκ Ζελντερλού. Ευχαριστώ. Τι ωραία που προφέρατε το όνομά μου. Δύο-τρεις παρατηρήσεις πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπε ο κύριος Πυρίνσκι. Να μην ξεχνάμε ότι μα ενδιαφέρουν οι αξιοπρεπεί θέσει εργασία που να έχουν και νόημα και ουσία. Να επιτρέπουν στου ανθρώπου να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν, να πραγματώσουν τα όνειρα και τι επιθυμίε του στη ζωή. Αυτού του είδου οι θέσει εργασία είναι οι πιο σημαντικέ. Τέτοιε αξιοπρεπεί θέσει εργασία απαιτούν και καλή εκπαίδευση. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το αγαθό τη παιδεία. Όταν μιλάμε για αξιοπρεπεί θέσει εργασία επίση, συμφωνώ με αυτό που είπε ο συνάδελφο πίσω μου, ο κ. Μπαρθ. Στι περισσότερε δημόσιε υπηρεσίε απασχόληση δεν έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία οι εργαζόμενοι για να καλύψουν όσου θέλουν στήριξη, ειδική στήριξη αλλά μπορούμε να έχουμε την προσφορά των μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων φορέων τη κοινωνία εδώ για να καλύψουμε αυτό το χάσμα. Στην Ιρλανδία, η κρατική υπηρεσία απασχόληση έχει τακτικές επαφές με τους φορείς στήριξης για άτομα με αναπηρίες για να είναι βέβαιοι ότι έχουν τη σωστή προσέγγιση και στη Φλάνδρα, στο Βέλγιο, στη δική μου την ε, περιοχή. Οι τοπικοί φορείς για την απασχόληση προβλέπουν στην δομή τους κάποιες φορές ένας άνθρωπος ε, από μη κυβερνητική οργάνωση συνήθως να προσφέρει στήριξη λόγω χάρη σε άτομα με αναπηρίες. Έτσι λοιπόν υπάρχει τρόπος να επιληθούν όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας κυρία Πρόεδρε για, την, για τον σχεδιασμό μια θέση εργασίας. Ε, είναι πολύ πετυχημένη η προσέγγιση, αλλά πώς να πείσουμε του εργοδότε. Ε, αυτό που πρέπει να ξεκινήσει κανεί είναι η επικοινωνία. Οι εργοδότες, οι κρατικέ αρχέ ε, απασχόληση, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει που στηρίζουν του διάφορου ανθρώπου, μιλούν διαφορετικέ γλώσσε και γι' αυτό πρέπει να έχουμε τόπου όπου όλοι συναντιόμαστε μεταξύ μα, με τι ίδιε εκφράσει, την ίδια ιδιόλεκτο και τρόπο που να συνεννόμαστε. Η δική μου οργάνωση συνεργάζεται με τους ανθρώπινους πόρους πολλών πολυεθνικών. Ξέρω ότι υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον δίκτυο από τον ILO, ε, business και disability, δηλαδή εταιρείε και αναπηρίες, ε, ώστε οι διαδικασίες πρόσληψης να γίνονται πιο ε, φιλικές προς τους χρήστες και πιο αποτελεσματικές. Αλλά το υπέρτατο είναι η επικοινωνία. Από εκεί πρέπει να ξεκινούμε. Γι' αυτό η εμπλοκή των εταίρων είναι πολύ σημαντική. και εκτός από Γενικός Γραμματέας της ESPD είμαι και ε, πρόεδρος μιας ε, επαγγελματικής ένωσης ε, απασχόλησης για ανθρώπου με αναπηρίες. Στο παρελθόν εκπαιδεύαμε, εκπαιδεύαμε του ανθρώπου συνεχώ. Και κάποιοι δεν έφευγαν ποτέ από την εκπαίδευση, από την κατάρτιση. Δεν έκαναν ποτέ αυτό το άλμα προς την αγορά εργασία. Τώρα τι κάνουμε, πηγαίνουμε και μιλάμε με τους εργοδότες τους ίδιου και τους λέμε πώς να εφαρμόσουν τα προγράμματα τα εκπαιδευτικά με τους συνεργάτες τους και το προσωπικό τους και αυτούς που ήδη εργάζονται στην εταιρεία. Δηλαδή να προβλέψουν νέες θέσεις εργασίας και δουλεύει αυτό. Είναι εφικτό. Το είπε και ένας από τους προηγούμενους ομιλητές. Ο κύριος Τόμπιν. Ναι, ίσως πολύ, δύο πολύ γρήγορα σχόλια. Το πρώτο είναι ότι πρέπει όντω να αναγνωρίσουμε ότι οι ενεργέ πολιτικέ απασχόλησει δεν είναι επανάκια. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα όπω οι συλλογικέ συμβάσει και διαπραγματεύσει, όπω ο κοινωνικό διάλογο. Το πλαίσιο εντό του οποίου όλα αυτά ε, αλληλεπιδρούν, η νομοθεσία προστασία τη εργασία, ε, οι άλλοι φορεί που ασχολούνται με την αγορά εργασία, η ελάχιστη μισθή και ούτω όλα αυτά πρέπει να ε, μελετηθούν από κοινού για να δούμε πώς αλληλεπιδρούν σε αυτούς που δεν έχουν κάποια δουλειά αλλά ως προς τις δεξιότητες τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο να προβλέψει κανείς ε, από το μέλλον. Βεβαίω το λέω αυτό αλλά πρέπει να πω ότι η ε, βελτίωση των δεξιοτήτων σε αυτούς που παραμένουν άνεργοι για πολύ καιρό είναι κάτι που φθήνει διαρκώς, ενώ οι δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας εξελίσσονται επίσης διαρκώς. Υπάρχει συνεχώς ένα χάσμα μεταξύ ζήτησης και προσφοράς και αυτό μπορεί πραγματικά να οξύνει τα πράγματα. Ναι, είναι πολύ σημαντική η κατάρτιση και η εκπαίδευση, αλλά πραγματικά αυτό που χρειαζόμαστε είναι να, είμαστε, να δράσουμε εγκαίρω, όσο το δυνατόν νωρίτερα, να είμαστε δραστήριοι και να έχουμε αποτελεσματικά ε, μέτρα, ώστε να δούμε ποια είναι η τελική στόχη που θέλουμε να πετύχουμε με τι πολιτικέ μα προ όλες τη οικονομία. Ε, Σα ευχαριστώ και ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας Απόντα που δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ και τους συντονιστές για την οργάνωση αυτής της ακρόασης. Ε, οι εισηγητές ήταν εξαιρετικοί με πολλές γνώσεις και ήταν ιδιαίτερα ενθουσιαστικό το να συζητάμε μαζί τους η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής μας 7 Δεκεμβρίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς και οι διερμηνείς σας ευχαριστούν για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε λοιπόν λέει η Πρόεδρος όλους. Γεια σας και καλή επάνωδο εύχομαι στους συγητές μας, τους προσκαλεσμένους μας. Ευχαριστώ. Γεια. Καλό απόγευμα.